Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε αμέσως με έναν πολύ απλό τίτλο. Διαπραγματεύσεις TTIP, Διατρεπτική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, αλλά περίπλοκο το θέμα. Να δούμε τι θα μας πει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Πέτρος Ουρνελής, υπεύθυνο τη ε, υπηρεσία για την πρόσβαση στην αγορά, την βιομηχανία, την ενέργεια και τι πρώτε Της τη DigiTrade στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Πρώτο ομιλητή θα είναι ο κύριο Χούμπαν, υπεύθυνο για τι σχέσει με τι Ηνωμένε Πολιτείε, τη DigiTrade στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Σα ευχαριστούμε που ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για τον 7ο γύρο των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτείων που έλαβαν χώρα στο Σέβι, στο Μερίλαντ από τις, 27, από τις 29 Σεπτεμβρίου στις 3 Οκτωβρίου του 2014. Όπως θα θυμάστε, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν επισήμως τον Ιούλιο του 2013. Ε, αυτός ήταν 7ο γύρος και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούνκερ, έχει εντοπίσει τις της TTIP ως μία από τις δέκα προτεραιότητες για την ε, νέα Επιτροπή που μόλις αναλάβε τα καθήκοντά της. Είναι σημαντικά σχετικά και τα αποτελέσματα των εκλογών ε, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ στις 4 ε, Οκτωβρίου. Όπως ξέρετε τον ε, έλεγχο της γερουσίας τον έχει πλέον ε, το κόμμα των ε, Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες αυτές εκλογές μέχρι την επόμενη επίσημη εκλογή του Αμερικανού Πρόεδρου. Αυτό μπορεί να επηρεάσει το μέλλον των διαπραγματεύσεων και μπορεί μάλιστα ο αντίκτυπος να είναι σοβαρός. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε την άποψή σας για το θέμα αυτό. εάν μπορούσατε να κάνετε την παρουσίασή σας σε 15 λεπτά, διότι μετά θα υπάρχουν και ερωτήσεις από τα μέλη και ίσως να είναι ακόμη πιο σημαντικό η συζήτηση που θα γίνει. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπεντ Λάγκε, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικού Εμπορίου. Και οι δικές σας παρατηρήσεις είναι πολύ κέρυες, διότι εσείς υγείστε τις αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά και βεβαίως και η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται πολύ για τη δική σας τοποθέτηση. Θέλουμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας ώστε όλοι να συντονιστούμε και να έχουμε κοινή προσπάθεια για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι σημαντικό βεβαίως και για το Ευρωκοινοβούλιο. Συνάδελφοι, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαι ακόμα και μέλος εδώ στην Επιτροπή Βιομηχανίας βέβαια και κατά τη διάρκεια της τελευταίας ε, εκλογικής περίοδου μπόρεσα να εργαστώ επ' αυτόν, αλλά αυτό καταδεικνύει ότι για μένα για την ε, δική μου κοινοβουλευτική επιτροπή και την Επιτροπή Βιομηχανίας συνδέονται πολύ στενά αυτά τα θέματα για την επανοβιομηχανοποίηση της Ευρώπης που θέλουμε να προαγάγουμε. Κατά τούτο λοιπόν αυτή η συμφωνία TTIP με τις ΗΠΑ είναι ένα σαφέστατο μέσο ώστε οι βιομηχανικές πιθανότητες ανάπτυξης στην Ευρώπη να βελτιωθούν. Και περί αυτού πρέπει να πρόκειται στα ουσιοδέστερα στοιχεία του ως εγχείρημα και στους 7 γύρους διαπραγματεύσεων εντωμεταξύ είδαμε ότι σε κάποιους τομείς πράγματι υπάρχουν δυνατότητες η βιομηχανική παραγωγή να ενδυναμωθεί στην Ευρώπη. Και έτσι λοιπόν η κατά μέσον όρων χαμηλοί τελωνιακοί δασμοί μπορούν να μειωθούν, αλλά πρέπει να δούμε πού υπάρχουν υψηλοί τελωνιακοί δασμοί και που παρακολύουν την πρόσβαση στην αγορά για επιχειρήσεις. Έχουμε ακόμα το φαινόμενο που για επιμέρους αυτοκίνητα, οχήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ 25% δασμός ε, εισπράτεται διότι δεν κατηγοριοποιούνται ως γιοταχή αλλά ως ε, γεωργικά οχήματα. Και σε πολλούς τομείς της τεχνικής, ε, των τεχνικών προδιαγραφών έχουμε παρόμοιες προδιαγραφές που οδηγούν σε παρόμοια αποτελέσματα όπως για παράδειγμα στο crash test δηλαδή ασφάλεια σε περίπτωση συγκρούσεων, όμως ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες εκάστοτε και κατά τούτο πιστεύω ότι και εδώ αξίζει τον κόπο να διαπραγματευτούμε με τη ΣΥΠΑ ώστε να υπάρξει ένα συνεκτικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο που θα συγκλίνουν οι προδιαγραφές και θα ενδυναμωθούν οι ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία έτσι. Ε, παρομοίως και σε άλλους τομείς των διαπραγματεύσεων υπάρχουν σαφέστατες δυνατότητες, τομεακά, κλαδικά συνάδελφοι, όπου η συνεργασία μπορεί να είναι ίσως κάπως πιο περιορισμένη διότι είναι διαφορετικά τα θέματα, οι προδιαγραφές τα χημικές, στις χημικές ουσίες. Καταλήξαμε στο REACH στην Ευρώπη. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στις ΗΠΑ όμως και υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες συνεργασίας και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό ως γεγονός. Συνολικά όμως υπάρχει ένα ευρύτατο πεδίο δυνατοτήτων συνεργασίας ώστε η επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης να ενταθεί, να ενισχυθεί και θα έπρεπε πραγματικά να κάνουμε χρήση αυτής της δυνατότητας και με παροχή υπηρεσιών που θα βρίσκεται κοντά στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Και φυσικά σκεφτήκαμε για ένα κεφάλαιο ενέργειας, ε, που η ενέργεια είναι, ας το πω έτσι, το λιγότερο ρυθμισμένο διεθνώς ε, ζήτημα και αξίζει τον κόπο να κάνουμε κάποιες προδιαγραφές στις οποίες θα καταλήξουμε ώστε να κατηγοριοποιηθούν τα καύσιμα όπως πρέπει μέσα σε ένα πλαίσιο συνεκτικό και να έχουμε ένα πρότυπο μέσα σε αυτή τη συμφωνία που πρέπει να αποσαφινιστεί καλύτερα όμως. Τώρα, όσον αφορά τώρα τις τηλεπικοινωνίες, πιστεύω ότι δεδομένων των αναγκών και για την ψηφιακή ανάπτυξη των επιχειρήσεων για το ψηφιακό μέλλον υπάρχουν σαφείς δυνατότητες ανάπτυξης του οικονομικού δυναμικού. Ωστόσο όμως από την άλλη πλευρά και εδώ πάλι ισχύει σε μεγάλο βαθμό αγαπητοί συνάδελφοι το θέμα της προστασίας δεδομένων που πρέπει να γίνεται σεβαστή προστασία των δεδομένων. Μια χαλήνοτη ροή δεδομένων σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο εκπροσωπεί τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και δεν τα αντανακλά και χωρίς ένα σωστό πλαίσιο ρύθμισης προστασίας των δεδομένων θα έχουμε κάποια όρια στα οποία θα προσκρούσουμε. Τώρα, πέρα από άλλες φοβι... όλες τις φοβίες ή επιφυλάξεις που με κριτικό πνεύμα πολλές φορές εκφράζονται, υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Και στην Επιτροπή Ανάπτυξης τίθεται πάλι η σαφέστατη προοπτική ότι σε στενή συνεργασία, όπως πρέπει, με την Επιτροπή Βιομηχανίας πρέπει να πορευθούμε στο μέλλον και να ε, προαγάγουμε θέματα. Και η συνεργασία αυτή αγαπητέ πρόεδρε κύριε Μπούζεκ μεταξύ μας είναι υποδειγματική μπορώ να πω. Ώστε πραγματικά από κοινού αυτό το πλοίο TTIP που είναι ένα μεγάλων διαστάσεων πλοίο να το φέρουμε σε αίσιο πέρα σε ένα ανασφαλή λιμένα με ρεαλιστικό πλαίσιο και κατεύθυνση. Και γι' αυτό ανήκει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια σε αυτό το εγχείρημα. Πιθανόν το, ε, η εντολή που πριν από δύο εβδομάδες ε, δημοσιοποιήθηκε με κάνει να πιστεύω ότι και με τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσουμε μεγαλύτερα πλαίσια διαφάνειας ώστε σε ένα επικοδομητικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών που θα διεξαγάγουμε να προχωρήσουμε σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλή συνεργασία που είχαμε και υπό αυτό το πνεύμα και την προοπτική ας συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Θα σας ζητήσω να τοποθετηθείτε και στο τέλος της συζήτησής μας και να ζητήσω τώρα από τους ε, ομιλητές μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταθούν σε κάποια ζητήματα που είναι πιο ενδιαφέροντα για τη δική μας την Επιτροπή, όπως τα θέματα των ρυθμίσεων, την ενέργεια και τις πρώτες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως, τα βλέπετε και στις ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Ποια είναι τα πλέον σημαντικά για μας. Θα έλεγα λοιπόν να ακολουθήσουμε την εξή σειρά. Ο κύριος Χάουερ να ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ πολύ και χαίρετε. Θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι ο Πέτρος στα δεξιά μου είναι ο υπεύθυνο για τις περιπλωτικές διαπραγματεύσεις. Εγώ ε, εργάζομαι από την γίδα του Ιγνάσιο που είναι ο, ε, ο πρώτος διαπραγματευτής, ο υπεύθυνος διαπραγματευτής. Να ξέρετε ότι, ξέρ, ότι καταλαβαίνουμε το πολιτικό ενδιαφέρον που έχουν και για το δικό σας σώμα οι σχετικές διαπραγματεύσεις. Και εφόσον ολοκληρωθούν μάλλον θα είναι η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που θα έχει ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο από τη θέση σε ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, κατανοούμε λοιπόν ότι θα πρέπει εδώ να συμπορευτούμε σε διαρκή διάλογο με την Επιτροπή ΙΝΤΑ και προκειμένου αυτά που λέμε και αυτά που προσπαθούμε να πετύχουμε να γίνονται κατανοητά και να τα συμμερίζεστε και εσείς. Είναι η τρίτη μέρα από την ανάληψη καθηκόντων του νέου μας επιτρόπου. Δεν μπορώ λοιπόν, σε, της νέας μας επιτρόπου, δεν μπορώ σε πολλά ε, να, να, πω τι θα γίνει και τι σκέφτεται, διότι ταξιδεύει ήδη στην, ε, α, ταξιδεύει προς την ε, από τη Σουηδία ε, για να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε. Τώρα, είναι σαφώς υπέρ της ε, ε, ελεύθερης αγοράς ως προς την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική, υπέρ των υψηλών προδιαγραφών προστασίας και της μεγαλύτερης διαφάνειας. Νομίζω θα τα δείτε εσείς και θα τα πει και στον πρόεδρο Λάγκε πολύ σύντομα, ώστε να βεβαιωθούμε ότι όλες αυτές οι προτεραιότητες θα εκφραστούν σωστά. Επίσης, την ακρόαση είπε ότι είναι υπέρ μιας νέας όθησης της διαπραγματεύσης TTIP, διότι τρόπον τεινά το 2014 οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο Βέβαια δεν πρέπει να υπερβάλλουμε, διότι υπήρχε και πολιτική μετάβαση εδώ στην Ευρώπη, που τώρα έχει πλέον ε, ολοκληρωθεί. Και υπήρχαν και οι χθεσινές εκλογές ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε λοιπόν να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το μήνα, εάν ε, καλά έχω καταλάβει, η Επίτροπος θα συνεννοηθεί με τους Ευρωπαίους ενδιαφερομένους με το θεσμικό σας όργανο, με το Συμβούλιο, με την κοινωνία των ε, πολιτών και τους εκπροσώπους της. Νομίζουμε ότι η πρώτη συνάντηση με τους Αμερικανούς στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων θα λάβει χώρα μόνον αφού έχει όλες αυτές τις συνομιλίες με τους ε, ενδιαφερομένους στην Ευρώπη. Όπως ξέρετε, ως προς τις διαπραγματεύσεις TTIP ξεκινήσαμε δημόσιες ε, διαβουλεύσεις και για το ISTS, το, κεφάλαιο, το εργαλείο αυτό που έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο επενδυτικό κεφάλαιο. Θα δούμε τώρα το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, πάρα πολλές όπως καταλαβαίνετε για δημόσιες διαβουλεύσεις. Πάνω από 1.500 απαντήσεις λάβαμε και θα ήθελε να παρουσιάσει η Επιτροπός μας τις απαντήσεις αυτές, την ε, συνεισφορά όλων στο κολέγιο των Επιτρόπων για να υπάρξει μετά και ο απαραίτητο διάλογο με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Μπορείτε λοιπόν να τα περιμένετε αυτά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ως προς τις Ηνωμένε Πολιτείες, χθες ε, ήταν οι εκλογές, η Γερουσία πλέον άλλαξε χέρια. Όλες οι προεδρίες των επιτροπών θα αλλάξουν από τον Ιανουάριο Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει πρώτα να δούμε τι προτεραιότητες θα θέσουν οι Ρεπουμπλικανοί που θα ελέγχουν το σώμα της Γερουσίας. Φαντάζομαι ότι στο Κογκρέσο και στη Γερουσία θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες ε, συνεννοήσεις ώστε οι Ρεπουμπλικανοί να συνεννοούνται με τους ομολόγους τους. Και θα περιμένουμε να δούμε και τις ε, ανάλογες μετακινήσεις στην ε, ηγεσία των δημοκρατικών στο Κογκρέσο. Οπότε μέσα στο πρώτο μισό του 2015 θα δούμε νομοσχέδια προς τον πρόεδρο από την εμπορική αρχή και βεβαίως και τις ανάλογες κινήσεις που προβλέπονται από το συνταγματικό σύστημα των ΗΠΑ, κάτι που ελπίζουμε ότι θα δώσει νέα όθηση στις διαπραγματεύσεις TTIP, διαπραγματεύσεις που παράλληλα διεξάγονται από αμερικανικές πλευράς και με ασιατικές χώρες. Το 2015 είναι κρίσιμη ε, χρονιά για τον Αμερικανό διαπραγματευτή, διότι συνειδητοποιεί ότι κάποια πράγματα θα ήθελε να ολοκληρωθούν προτού η χώρα ε, περάσει σε φάση προεκλογική, το 2016 δηλαδή. Υπ' αυτήν την έννοια το 2015 για τις ΗΠΑ είναι μια χρονιά σημαντική. Θέλει μαζί με τους Ευρωπαίους να προχωρήσει ε, ώστε οι διαπραγματεύσεις TTIP να μπουν σε μια τροχιά προς την επιτυχία. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε κάποιο χρονικό ορίζοντα και κάποια αντικείμενα προς εξετάση. Νομίζω ότι εσείς μπορείτε να ηρεμήσετε. Έχετε πέντε χρόνια μπροστά σας. Ε, είσαστε κι εσείς κάποιοι εντελώς νέοι, όπως και η Επίτροπος ε, εν μέρη, οπότε θα ε, δούμε τι θα γίνει και το 2015 και το 2016. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της θητείας σας θα φτάσει στα χέρια σας σίγουρα η συμφωνία αυτή για να αποφασίσετε. Πολύ σύντομα και για να ολοκληρώσω πρωτού δώσω το λόγο στον συνάδελφο Πέτρο ε, να πω που έχουμε φτάσει στις διαπραγματεύσεις αυτές καθεαυτές. Ε, έχουμε ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο, ε, είχαμε πέντε γύρους. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι τα πράγματα δεν έχουν πάει άσχημα για δουλειά ενός χρόνου. Στους περισσότερους τομείς όπου υπάρχει διαπραγμάτευση προχωρούμε με κοινά κείμενα, δηλαδή ένα κείμενο με στήλε όπου υπάρχουν, ε, υπάρχει μάλλον ένα κοινό κείμενο στη μέση και όπου υπάρχουν διαφωνίες σημαίνονται σε δύο διαφορετικές στήλε. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν labor και environment, εργασία και περιβάλλον. Εκεί υπάρχουν ε, κάποιες αποκλήσεις, εκεί δεν υπάρχει ακόμα κοινό κείμενο. Για κάποια από τα θέματα που ανέφερε ο κύριος Λάγκε επίση είναι κεντρική σημασία για τις δημοκρατεύσεις, δεν έχει ακόμα συνταχθεί το σχετικό κείμενο. Για το κομμάτι της πρόσβασης στην αγορά ούτε αυτά έχουν ολοκληρωθεί. Πρέπει να δούμε πώς θα απελευθερώσουμε την αγορά μας σε τομείς που ακόμη είναι προστατευόμενες. Υπάρχει ακόμη αρκετός προστατευτισμός ε, και αυτό πρέπει να γίνει με παραχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι προφανές για διαπραγματεύσεις μιλάμε. Και μετά νέους κανόνες. Οι διαπραγματεύσεις θέλουν να καταλήξουμε και σε ένα σύνολο κανόνων που κάποια στιγμή θα γίνουν ένα μοντέλο ένα ορόσημο που θα μπορούσε να αντιγραφεί και για άλλες ε, εμπορικέ συμφωνίες ή δυνατόν κιόλα για τον ΠΟΕ στη Γενέβη. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν κάποια διαφορετικά θέματα, την πρόσβαση στην αγορά, την ρυθμιστική συνεργασία, χωρίς να μειωθούν οι προδιαγραφές προστασίας και η θέσπιση νέων κανόνων σε κάποιου τομείς όπου ακόμη δεν υπάρχουν. Αυτά είναι μεσοπρόθεσμοι στόχοι στρατηγική σημασία. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό που έδωσε ο κ. Λάγκε για τα δεδομένα και οι διαφορετικοί τρόποι κατά τους οποίους αποθηκεύονται, ανταλλάσσονται στις σύγχρονε οικονομίες τα δεδομένα. Ασχολούμαστε και με τα επίπεδα απορρίτου εμπιστευτικότητας και αυτά μπορεί να ε, επηρεαστούν. Ε, φυσικά δεν θέλουμε να μειώσουμε πουθενά το επίπεδο προστασίας. Η εμπιστευτικότητα εξετάζεται και αλλού βάσει της νομοθεσίας που έχετε εγκρίνει κι εσείς, αλλά ως προς την ε, απελευθέρωση του άνοιγμα της αγοράς. Αυτό προφανώς ενδιαφέρει τους διαπραγματευτές εμπορικών ε, υποθέσεων και βεβαίω επηρεάζει, έχει μεγάλη σημασία και για την οικονομία εντό τη οποία ζούμε. Με αυτά έχω ολοκληρώσει να δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον Πέτρο. Yes, thank you very much, uh, Chairman. Good afternoon. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μετά την ε, εισήγηση του συναδέλφου, εγώ θα μπορούσα να είμαι πιο συγκεκριμένος από τα πιο τεχνικά ζητήματα όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά τις πρώτες ε, ύλες, όσον αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις. Μια από αυτό το κομμάτι είναι εγώ. Πρόκειται για κάποια τέτοια υλικά που είναι ζήτημα μεγάλο του 21ου αιώνα, είναι μια πρόκληση όλο ένα και πιο μεγάλη, αλλά είναι κάτι το οποίο, όπως είπε ο πρόεδρος Λάγκε, ε, που ακόμη δεν έχει καλυφθεί όπως πρέπει από τους διεθνείς κανόνες, από τους, τις διατάξεις του ΠΟΕ, ε, οπότε υπάρχουν εδώ πέρα σημαντικά κενά και επομένως οι σημερινές υπάρχουσες διατάξεις δεν μας καλύπτουν. Και για αυτόν τον λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τις διαπραγματεύσεις TTIP ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιους κανόνες παγκόσμιους και έτσι να έχουμε έναν αριθμό διατάξεων που να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους εμπορευόμενους σε αυτόν τον τομέα. Υποβάλαμε πριν από ένα χρόνο τις προτάσεις μας προς τις είπα, για κάποιες ε, διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στο κεφάλαιο για ενέργεια και πρώτες ύλες με αυτές τις ε, διατάξεις προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων. Τις εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις για δραστηριότητες της για διαφάνεια, για αποφυγή δυσμενών διακρίνων, για κάποιες ε, ε, πρακτικές καθορισμού των τιμών, σε σχέση με την, ε, κάποιες πρακτικές μάλλον διτής τιμολόγησης όσον αφορά τις ε, προβλεπόμενες νομοθετικά τιμές όπου υπάρχουν σε κάποιες χώρες, κάποιους διατίμηση δηλαδή και επίσης ε, είπαμε για την απαγόρευση μονοπωλίων, εξαγωγών, για το δικαίωμα πρόσβασης τρίτου όσον αφορά τις ε, μεταφορικές υποδομές, φερειπίν τα δίκτυα ηλεκτροδότησης ή τους ε, αγωγούς. Σημαντικά αυτά για πολλές χώρες και επίσης κάποια άλλα ζητήματα ασφαλείας ε, όσον αφορά επίσης κάποιες κινήσεις, κάποιες συναλλαγές που αφορούσαν, αφορούν υπεράκτιες ε, επικράτειες. Οπότε επίσης τώρα είχαμε και το σημαντικό ζήτημα του πώς θα αρθούν οι περιορισμοί οι Αμερικανικοί για το αργό πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο. Πολύ σημαντικός στόχος για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την Ένωση. Πέραν επομένω αυτών των στοιχείων για τα ε, ορυκτά καύσιμα, πέραν του και κεκτημένο που υπάρχει. Είχαμε και κάποια ζητήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ένας κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται και πρόκειται να αποσχολήσει τις διαπραγματεύσεις τους επόμενους γύρους. Τώρα, οι Ηνωμένε Πολιτείε ακόμη δεν προχώρησε μια πολιτική απόφαση όσον αφορά το να καλυφθεί η υπόθεση ενέργεια και πρόταση της από κάποιο κεφάλαιο και έτσι να έρθουν και οι περιορισμοί όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση περιορισμοί των εξαγωγών και έτσι δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημη απάντηση στην πρότασή μας. Και εξαγωγές τώρα υγροποιημένου φυσικού αερίου, η θέση τους είναι ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιληθεί αφού ολοκληρωθεί ε, το TTIP με κάποια συμφωνία ελευθερών εμπορίου. Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις ΗΠΑ αυτόματη χορήγηση άδειων και Αυτό βέβαια σημαίνει μονόπλευρη και μονομερή λήψη απόφασης. Δεν πρόκειται για κάποια δέσμευση της συμφωνίας. Πολύ σημαντικό αυτό να το τονίσουμε. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το να θεωρήσουμε αναλογικά και στις εξαγωγές του αργού πετρελαίου. Βεβαίως και το θέμα έχει σημασία γεωστατηγική και αυτό επίσης έχει τονιστεί και ανταγωνιστικότητα, στόχοι, συστημική. Ε, εμείς εξηγήσαμε σε πολιτικό επίπεδο αυτό το οποίο ζητούμε. Ταξιδέψε και εκεί ο πρώην Επίτροπος ο κ. Ντεχίχ το Σεπτέμβριο και όπως ακούσατε και στην ακρόαση η Επίτροπος Μάλιστον ε, αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα. Περιμένουμε επομένως την απάντηση των Αμερικανών. Συνεχίζουμε το έργο μας, τις επαφές σε διάφορους γύρους, σε διάφορα θέματα, όλα αυτά περιέχονται στην ε, γραφό μας. Πάμε για τον 7ο γύρο, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση τρίτων στις ε, μεταφορικές υποδομές, για τα θέματα διαμετακόμισης και επίσης ε, συζητήσαμε και τις ε, αναθεωρημένες διαδικασίες για τις άδειε εξαγωγών. Θέλουμε να δούμε τι κοινά σημεία έχουμε, οι μεν και οι δε στην ομοθεσία μας, να δούμε οι δημιουργικές αρχές, τι τεχνικές δεν αντιμετωπίζουν, να δούμε ο πλευράς Αμερικανών τι θέλουν, τι σκοπεύουν, αλλά τέλος πάντων περιμένουμε την επίσημη απάντηση ακόμη. Για τον επόμενο γύρο, επαναλαμβάνω ενανεμόνη τη απαντησεώ του. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει για να νιώσουμε τι πηγέ ενέργεια και για ζητήματα ενεργειακής αποτελεσματικότητας. Και άλλα θέματα είχαμε, αλλά ακόμα δεν βρήκε ο χρόνος να συζητηθούν. Έτσι έχει η κατάσταση των πραγμάτων προς το παρόν. Βεβαίως και ελπίζουμε ότι σύντομα θα απαντήσουν, είπα, στις προτάσεις μας. Και έτσι θα είμαστε εις θέση να συζητήσουμε πέραν των τεχνικών ζητημάτων σε κάποια αυθεντικά διαπραγματευτικά ζητήματα. Ευχαριστούμε του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Πρόεδρο. Και τώρα, οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων α πάρουν το λόγο. Συνάδελφοι, δύο λεπτά παρακαλώ. Μέσα με την πρώτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ενημέρωση. Κάποιες λίγες παρατηρήσεις και ερωτήσεις μόνο. Δημόσιες προμήθειες. Το Σεπτέμβριο εμείς σε αυτή την όχθη του Ατλαντικού αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε και το Μαυροβούνιο και τη Σερβία στις ρυθμίσεις αυτές. Αυτό δημιουργεί το ερώτημα πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά με την προσέγγιση των ΙΠΑ σε σχέση με αυτό το θέμα αν μια τέτοια συμφωνία μπορέσει να επιτευχθεί με τις ΗΠΑ, πού αυτές οι τρίτες χώρες θα μπορούσαν να συσχετιστούν μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων για τις ε, δημόσιες προμήθειες. Τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βλέπω στην έκθεση για την 7η συνάντηση αναφέρεται ότι η πλευρά των ΗΠΑ έθιξε κάποια θέματα για τα θέματα συμμετοχής των ΜΜΕ στις ε, διαδικασίες συμμετοχής, αξιολόγησης κτλ. Πώς απαντά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Ποια ήταν τα αίτια, ήταν ε, μια κριτική παρατήρηση, ποια ήταν, ποιο ήταν το περιεχόμενο, η ουσία επ' αυτού είναι όσο πιο θα έλεγα ουδέτερες και αδρανείς ε, οι παρατηρήσεις και τα στοιχεία που μας δίνονται που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με αυτά τα θέματα. Τρίτον, επιχορηγήσεις, γεωργία, επιδοτήσεις, ε, βαμβάκι. Κλινικά έχει εξηγιανθεί το θέμα από τα όσα μας υποβάλλονται ως έγγραφα με στοιχεία για αυτά τα ζητήματα. Αλλά για τη συζήτηση και σύντομα επισημένοντας αυτά που ανέφερε ο πρώτος ομιλητής, αυτό είναι το στοιχείο για όλες τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που ε, ελπίζουμε να είναι, να, ε, είναι μακρόβιες και να είναι σε ένα ισχυρό θεμέλιο. Αλλά τι γίνεται σε σχέση με άλλα τρίτα μέρη στην παγκόσμια κλίμακα και ποια είναι η αντίδραση σε σχέση με αυτή την μελλοντική συμφωνία όπως ελπίζουμε που θα συναυθεί σε σχέση με αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Λίνα παρακαλώ. My Σειρά μου. Λυπάμαι λοιπόν πολύ που καθυστέρησα. Κυρία Μίλναρ, Μλίναρ, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που, καθυ... που χρησιμοποιώ τον χρόνο σας. Δύο συγκεκριμένες παρατηρήσεις έχω. Πρώτον, προέρχομαι από την Αυστρία, που είναι μια χώρα που έχει πολλές επιφυλάξεις σε σχέση με αυτά τα θέματα, όπως θα γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στην αίθουσα. Εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτής της συμφωνίας και είμαι πεισμένη ότι το εμπόριο γενικά είναι η βάση της δημιουργίας πλούτου γενικά. Οι ερωτήσεις μου προς εμάς λοιπόν τώρα είναι αφορούν δύο θέματα. Πρώτα, βρισκόμαστε τώρα στη φάση του να προχωρήσουμε προς την αποδοχή του ΣΥΤΑ. Το ΣΥΤΑ πώς θεωρείτε εσείς ότι συνδέεται με, την, με τη συμφωνία αυτή. Αν περάσει το ΣΥΤΑ τότε θα έχουμε καλύτερη πιθανότητα προοπτική να έχουμε μια καλή ε, θέση κίνησης για την TTIP. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το ζήτημα των εθνικών κοινοβουλίων που και αυτά θα πρέπει να επικυρώσουν την τίτη. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού. Ευχαριστώ. Ε, ε, Σε ευχαριστώ κύριο Ετσενίκε παρακαλώ, επόμενος ομιλητής. Ετσενίκε. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Συνάδελφοι. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες ε, πρόσφατα και μία από το Πανεπιστήμιο Ταφτς που την έχω εγώ στα χέρια μου, στο τραπέζι μου. Οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν ότι οι επιπτώσεις όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπογράψει την TTIP θα είναι αμεσότατες ε, όσον αφορά την απασχόληση και το ποσοστό hm, όσον αφορά τα έσοδα που θα προέρχονται από την εργασία σε σχέση με τα κέρδη και έσοδα από το κεφάλαιο, οικολογικές επιπτώσεις και τα συναφή. Επίσης οι ΜΜΕ δεν θα μπορέσουν να υποφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Μάλλον το αντίθετο θα συμβεί. Και λένε και ακόμα ότι υπό τους όρους του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δεν θα είναι πολύ καλές οι προοπτικές. Τούτων λεχθέντων γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές θα υποφεληθούν από την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Η κύρια ερώτησή μου λοιπόν είναι τι θα γίνει με τους πολίτες της Ευρώπης, πώς θα υποφεληθούν και οι μικρές, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ευρωπαϊκές, ποιες επιπτώσεις θα υποστούν, πώς θα υποφεληθούν. Ευχαριστώ. Μπορέλη. Κύριε Μπορέλη. Τον τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε δόθηκε έμφαση και από τις δύο διαπραγματευτικές πλευρές την ανάγκη να συμμετάσχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο στη διαδικασία των διαβουλεύσεων ώστε να γίνουν γνωστές και οι πραγματικές τους ανάγκες. Ανεξάρτητες μελέτες, όλο ένα και πιο περισσότερες, δείχνουν πως οι ελεύθερες συναλλαγές με τις Ηνωμένε Πολιτείε μπορεί να, ε, ε, να προκαλέσει σοβαρή μείωση του ενδοκινοτικού εμπορίου για τις επιχειρήσεις αυτές λοιπόν, ιδίω τις μικρές, πώς θα είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Τι ε, στοιχεία υπάρχουν ε, για το πώς θα επιδράσει η Συμφωνία TTIP στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τι θα γίνει εφόσον οι εμπορικές ροές αλλάξουν κατεύθυνση σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, πώς θα συμμετάσχουν ενεργά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις διαπραγματεύσεις. Βάσει και της παρατήρησής σας ότι το εργαλείο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει χρησιμοποιήσει ως ω τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται ότι δεν ε, είναι αποτελεσματικό και σκόπιμο για τους σκοπούς αυτή της συμφωνία. Για το STS, λόγω χάρη, έχετε καταγράψει μια πολύ χαμηλή συμμετοχή. Όχι γιατί το θέμα δεν θεωρείται κέριο, αλλά γιατί αντιθέτω οι επιχειρήσει, ιδίω οι μικρομεσαίε, δεν ε, έχουν γνώση του θέματο. Πώ αξιολογούνται τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκίνησε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για την διαφάνεια των διαπραγματεύσεων TTIP που ολοκληρώθηκαν φέτο τον Οκτώβριο του 2014. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ίσως θα θέλατε να απαντήσετε σε μια πρώτη φάση. Ίσως να είναι καλύτερα έτσι. για τις ερωτήσεις του κυρίου Μέσας με δημόσιες προμήθειες. Σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ο σκοπός είναι να υπάρχουν αμοιβαία ωφέλη. Βασική αρχή είναι να ωφελούνται και οι δύο πλευρές και βεβαίως δεν, να μην ωφελούνται όσοι δεν είναι μέρη της συμφωνίας. Ε, είναι και συνήθεις κανόνες που ισχύουν στον ΠΟΕΟ... που οφέλη πρέπει να προσφέρονται προς όλους. Ό,τι δίνουμε στους Αμερικανούς μας δίνουν και εκείνοι στα πλαίσια του TTIP. Αλλά αυτό αφορά τις δύο πλευρές αυτής της συμφωνίας. Και θα ισχύσει κάτι τέτοιο και για τις δημόσιες προμήθειες, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επειδή πολλοί έθιξαν το θέμα αυτό, και είπατε ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι η συμφωνία θα ωφελήσει τις πολυεθνικές, τις μεγάλες εταιρείες που έχουν ούτως ή άλλως βρει το δρόμο τους από την ε, άλλη πλευρά του Ατλαντικού και λιγότερο τις μικρομεσαίες. Νομίζω από την αμερικανική πλευρά οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι συνολικά το μεγαλύτερο όγκο του εμπορίου τον καλύπτουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αν τα δείτε από μακροοικονομική σκοπιά. Είναι μικρό το ποσοστό των μικρομεσαίων όμως που εξάγουν και εισάγουν. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης εδώ στο ε, επίπεδο των μικρομεσαίων εάν απλοποιηθεί το διεθνές εμπόριο και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί κανείς είναι λιγότερο επαχθείς. Μέσα από αυτές τις διαπραγματεύσεις λοιπόν αναζητούμε μηχανισμούς για να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος, το άχθος για τις ε, μικρές αυτές επιχειρήσεις, αλλά να διατηρήσουμε τα επίπεδα προστασίας που έχουμε μεν και ιδέ στις κοινωνίες μας, στις αγορές μας, που κάποιες φορές διαφέρουν βέβαια. Η ε, τέχνη όλοι λοιπόν και ο σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διατηρηθούν μεν οι διαφορές, αλλά όχι όταν υπάρχουν μόνο για λόγους γραφειοκρατικούς, ε, τεχνικούς και δεν έχουν κάποια λογική. Λόγω χάρη τα crash test για τα οχήματα ή τις απαιτήσει για τις ζώνες ασφαλείας που είναι διαφορετικές ε, για τα γιοταχή. Αυτά έχουμε δει ότι δεν έχουν δραματικές διαφορές τα τελευταία 40 χρόνια. ή αυτοκινητοβιομηχανίες λοιπόν πρέπει να συμμορφώνονται με δύο διαφορετικές νομοθεσίες. Αυτό έχει σοβαρό κόστος και τελικά δεν κάνει κανένα ούτε πιο χαρούμενο ούτε πιο ασφαλή. Για αυτού του είδου τους κανόνες θέλουμε να μειώσουμε το άχθο. Ε, εφόσον όλα τα υπόλοιπα διατηρηθούν ε, όμοια, οι πρώτοι που θα ωφεληθούν είναι οι μικρές επιχειρήσεις, διότι οι μεγάλες ούτως ή άλλως έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τις υπάρχουσες, τους υπάρχοντες περιορισμούς. Πρέπει λοιπόν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρουν το δρόμο τους προς την Αμερικανική αγορά. Αλλά η General Electric λόγω χάρη ξέρει πώς να έρθει ω την Ευρωπαϊκή αγορά και η Siemens ξέρει πώς να πάει στην Αμερικανική. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει μια αλληλεπίδραση στο ε, διμερές αυτό εμπόριο που να είναι απλούστερη και να αμφεληθούν οι μικροί παράγοντες της οικονομίας. Για την γεωργία, οι επιδοτήσεις δεν είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων σε αυτή τη συμφωνία οι επιδοτήσεις είναι κάτι που μπορείτε να διπλωματευτείτε μόνο με όλους παγκοσμίω ε, στον, ε, στο παγκοσμίο προσκήνιο. Δεν μπορεί κανείς να πει θα αλλάξω την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική, μόνο αν αλλάξουν και οι Αμερικανοί κάτι στη δική του, στο δικό τους νόμο περί Γεωργίας, στο Farm Bill. Ε, πρέπει τα επίπεδα των επιδοτήσεων να κατέβουν παντού συντονισμένα σε όλες τις αγορές ταυτοχρόνως. Ε, για τι επιδοτήσει λοιπόν όχι, αλλά η απάντηση για την πρόσβαση στην αγορά, η απάντηση είναι και πάλι ναι. Ε, θα δώσουμε ε, διόδου πρόσβαση στην αγροτική μα αγορά, στην αγορά τροφίμων στι ΗΠΑ και το ίδιο ελπίζουμε και αναμένουμε να πάρουμε κι εμεί. Πρόσβαση στην αγορά των Αμερικανών. Είμαστε άλλωστε ένα από του μεγαλύτερου εξαγωγεί γεωργικών προϊόντων προ τι ΗΠΑ. Να σκεφτούμε λοιπόν ότι δεν έχουμε μόνο ε, ανάγκη να υπερασπιστούμε τη δική μα γεωργία, περισσότερο εξάγουμε παρά εισάγουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δείτε τι θέσει απασχόληση θα μπορούσαν να δημιουργηθούν. Υψηλή ποιότητα για τα τελικά προϊόντα. Ε, με τεράστια κέρδη μπροστά μα. Ιδίω για την πρόθεση προϊόντων με γεωγραφική προστατευόμενη με γεωγραφικέ ενδείξει και προστατευόμενη προέλευση θα μπορούσαν να φτάσουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτά θα ωφελήσουν του μικρού παραγωγού και όχι τι μεγάλε πολυεθνικέ. Για τη σχέση των διαπραγματεύσεων TTIP και τι τρίτε χώρε, όλε οι οικονομικέ μελέτε δείχνουν ότι οι τρίτε χώρε θα είναι οι πρώτοι που θα ωφεληθούν ακόμη και αν είναι μια προτιμησιακή συμφωνία αυτή. Δηλαδή η μείωση των επιπέδων προστασία αφορά μόνο τι δύο πλευρέ τη συμφωνία. Οι τρίτε χώρε θα ωφεληθούν, όπω ωφελήθηκαν και από την ενιαία αγορά όταν δημιουργήθηκε το τη δεκαετία του 80. Όλοι μίλησαν για την ε, Fortis Europe. Ε, θα το θυμάστε όσοι είστε μεγαλύτεροι. Για θυμηθείτε τι γινόταν τότε όταν ε, ε, κάποιο ήθελε να εξάγει προ την Ευρώπη, είχε πλέον μία προδιαγραφή κοινή να ε, σεβαστεί. Και έτσι μπορούσε να πουλήσει τα προϊόντα του σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτόχρονα. Άρα η συμφωνία αυτή θα δείξει σε ποια σημεία συμφωνούμε και σε κάποια σίγουρα θα διαφωνούμε. Αλλά όπου συμφωνούμε, με κοινέ προδιαγραφέ που θα ωφελήσουν και του ΜΕΝ και του ΔΕ, κατ' επέκταση θα ωφεληθούν και τρίτε χώρε. Για την κυρία Μλίνεν. Ε, έχουμε γνώση των όσων συμβαίνουν ε, στην Αυστρία και εδώ θα ζητούμε τη βοήθειά σας. Και σε κάποια άλλα κρατημέλη ξέρουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες. Ε, είναι μια ε, ένα θέμα συζήτησης που έχει λάβει μεγάλη προβολή. Δεν το περίμενα αυτό ως διαπραγματευτής. Αλλά εξηγήστε μας εσείς τι είναι για τους ψηφοφόρους σας η Συμφωνία TTIP. Και εφόσον δεν γνωρίζουν, εξηγήστε τους θα πρέπει να τους δώσετε κίνητρα, να τους το ε, κάνετε σαφές. Είναι ένα θέμα που έγινε πολύ δημοφιλές και θα πρέπει όλοι να αποκτήσουμε τις... Ε, σχετικέ γνώσεις. γνώσει. η σφαιρική και σε βάθος Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών, η ΣΥΤΑ, είναι ε, ένα μοντέλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη Συμφωνία TTIP. Δεν σημαίνει όμως ότι τα πράγματα θα τα κάνουμε ακριβώ ίδια. Ε, Η συμφωνία, η σφαιρική και σε βάθος συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών είναι μια συμφωνία που είναι από τις πιο σύγχρονες, τις πιο πρόσφατες που έχουμε ποτέ συνάψει. Πριν από δίμηνο συμφωνήθηκε, οπότε δείχνει το καλύτερο επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε σε σχέση με τι εμπορικέ μα προδιαγραφέ και δείχνει το δρόμο για του κανόνε που θέλαμε να προβλέψουμε. Για την όλη συλλογιστική λοιπόν των δημοκρατήσεων TTIP είναι ότι δεν Προσπαθούμε απλώς να ε, αξιοποιήσουμε την άκρατη παγκοσμιοποίηση, αλλά να προβλέψουμε και ένα σύνολο κανόνων για να υπάρχει ε, ελεύθερη αγορά, ένα ανοιχτό σύστημα προσφοράς και ζήτησης. Για την ανάμειξη ε, στη γενική διεύθυνσή μας, αυτό που λέμε είναι ότι όταν φτάσουμε σε αυτή τη γέφυρα θα την περάσουμε τότε. Δεν θα προτρέξουμε. Δηλαδή, θα δούμε ανάλογα με τις κανόνες που θα προβλέπονται στη συμφωνία και το πώς ορίζονται ε, από τη συνθήκη, θα δούμε τι θα κάνουμε τότε. Καταλαβαίνετε όμως ότι σε μια συμφωνία τέτοιας σημασίας θα περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα. Μπορεί να χρειαστεί να κυρώσουν τα εθνικά κοινοβούλια, το έχει πει κάποιος αυτό. Αλλά σκεφτείτε κι εσείς τι θα κάνετε το Ευρωκοινοβούλιο. Θα θελήσετε να πάνε τα πράγματα αυτά να φτάσει η συμφωνία στο Εθνικά Κοινοβούλια. Θα θελήσατε την ανάπτυξη της εμπορικής μας πολιτικής. Ε, Αλλαγέ στη συνθήκη έχουν γίνει και για άλλους λόγους. Εδώ έχουμε πολύ ε, σημαντικά θέματα μπροστά μας που και εσάς είναι ρόλο σας να τα σκεφτείτε. Όταν ήμουν υπάλληλο στα νιάτα μου, το Συμβούλιο ήταν το περιβάλλον που περιμέναμε να πάρουμε έγκριση για να προχωρήσουμε. Τώρα ε, είναι και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Για σκεφτείτε αν χωράνε σε αυτό το μοντέλο και τα Εθνικά Κοινοβούλια, διότι όσο πιο πολλά επίπεδα πρόοδου έγκρισης ε, για να προχωρήσει ένα θέμα προβλέψετε, τόσο πιο αργά θα πάμε. Η αν όμω το κάνουμε αυτό, οι Αμερικανοί θα πούν θα ψηφίσουμε και εμεί τη συμφωνία, αφού ψηφίσουν και τα 28 κράτη-μέλη. Για σκεφτείτε το λοιπόν, σκεφτείτε πόσο αξίζει τον κόπο. Για τι ερωτήσει τώρα για τι μικρομεσαίε νομίζω προσπάθησα να απαντήσω, αλλά και για του πολίτε. Σκεφτόμαστε και άλλε πτυχέ τη συμφωνία που απευθεία ε, ενδιαφέρουν του ε, πολίτε όλων των ηλικιών. Για την κινητικότητα, πώ μπορούμε να διευκολύνουμε τους εργαζομένους να πάνε στην άλλη αγορά με επιταχυμένες διαδικασίες ή πώς θα καλύψουμε τους νεότερους για τη διαφάνεια και πάλι το είπα και στην εισαγωγή μου η Επίτροπος θα έρθει που να είναι με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες νομίζω έχει κάποιες προτάσεις να κάνει θα τα συγκεκριμένει πρώτα με τον κύριο Λάγκε και μετά θα τα δείτε Ευχαριστούμε πολύ κυρία Έλνστα Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ προέρχομαι από μια περιφέρεια από την Ανατολική Γερμανία όπου η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει μεταξύ 10 και 15 απασχολούμενους. Είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως τις αποκαλούμε. Ή θα μπορούσαμε να τις αποκαλέσουμε μικροεπιχειρήσεις από πλευράς των ενώσεων και συλλόγων μεσαίων επιχειρήσεων υπάρχει μια ολόκληρη σειρά διεκδικήσεων και θεμάτων ως απαιτήσει για την TTIP, γιατί μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις οι διατάξεις αυτής της συμφωνίας για τις μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά που μας εκθέσατε δεν υπάρχουν καθόλου. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα έχουν ποτέ κάποια ευκαιρία όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν τελείως άλλες διαστάσεις ε, όπως τι είπα να κάνουν μεγάλα, μεγάλες συμφωνίες και να πολλούν πολλά οχήματα. Το θέμα των μικρών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντικό. Κάτι θα ήθελα να μου πείτε περισσότερο. Όχι μόνο για αυτές που υπάρχουν στην Ανατολική Γερμανία σήμερα, αλλά για αυτές που υπάρχουν και σε άλλα κράτη. Για μας είναι αδιαμφισβήτητο μια TTIP χωρίς συγκεκριμένες διατάξεις για την προστασία δεδομένων <clears throat> δεν επαρκεί. Πρέπει κάτι να γίνει για την προστασία των δεδομένων. Επίσης πείτε μου για την Global Development Environment Institute στο 15.3 όπου μια ολόκληρη σειρά σαφών μειονεκτημάτων απορρέων που μέσω της TTIP θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους, τους απασχολούμενους. Αλλά συγκεκριμένα χειροπιαστά τώρα, όχι γενικόλογα, να απαντήσετε ευχαριστώ. Καλίντς παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όρος διαφάνεια πραγματικά πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να τον σκεφτούμε, διότι είναι μια σαφής κατάσταση στην οποία καταλήγουμε όλοι σε σχέση με το ΕΛΚ είμαστε απόλυτα υποστηρίζουμε και είμαστε οπαδοί της TTIP. Είναι μια μεγαλόπνοη ιδέα σίγουρα. Τώρα έχουμε μια συζήτηση για θέματα που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση και δεν γνωρίζουμε τίποτα για τα διαδικαστικά και αυτό είναι κάπως ένα πρόβλημα. Κατανοώ φυσικά το ότι έχουμε διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις είναι διαπραγματεύσεις. Παρ' όλα αυτά ενδιαφέρον θα ήταν να μπορέσουμε να κατανοήσουμε στον τομέα των ενεργειακών, της ενέργειας και των πρώτων υλών τι γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια κοινή ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων ενέργειας, ενεργειακών προϊόντων. Είναι στόχος να το καταφέρουμε να το πετύχουμε. Στις διαπραγματεύσεις μας με τη ΣΥΠΑ αυτό διαδραματίζει κάποιο ρόλο. Ποια θέματα τίθενται π.χ. για τους Αμερικανούς που να μην ικανοποιούνται με αυτά. Ποια θέματα τίθενται για τους, απέναντι στους Ευρωπαίους τα οποία δεν τους ικανοποιούν και ποια θέματα δεν θέτουν προβλήματα σε αυτόν τον τομέα. Και μια δεν έχουμε μια τέτοια κοινή αγορά. Αυτό διαδραματίζει ή όχι ένα ρόλο. Πρέπει να το κατανοήσουμε και να δούμε τι γίνεται. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά ένας έσχιστος τρόπος να εργάζεται κανείς με αυτόν τον τρόπο υπό το πρίσμα του Κοινοβουλίου. Γιατί πράγμα μπορεί να κάνει κανείς λόγο μπορώ να κάνω λόγο εγώ στους ψηφοφόρους μου για μια ιδέα, ιδέα υπό εφαρμογή προς εφαρμογή, όπως αυτά που προτείνονται εδώ. Θέλω να κατανοήσω περί τίνος γίνεται λόγος εδώ, γιατί πράγμα συζητάμε. Συγκεκριμένα, ενέργεια, πρώτες ύλες. Πείτε μου, τι γίνεται σχετικά. Ποια είναι τα θέματα και διαδικασίες. Πώς όλα αυτά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την απουσία κοινή αγοράς για αυτά διαδραματίζει ρόλο ή όχι. Ε, Λόπες Μπερνέο. Λόπες Μπερνέο παρακαλώ τώρα. Μάλιστα, καλό σας απόγευμα σε όλες και όλους. Δεν συμφωνούμε ούτε επί της ουσίας, ούτε με τους τρόπους και διατυπώσεις για αυτή την πιθανή συμφωνία. Για τους τρόπους και διαφωνία και διαδικασίες, διότι παραμένουν θέματα λομπίστων που εκπροσωπούν συμφέροντα πολυεθνικών. Αν δεν υπάρχει κάτι να αποκρύψετε, να δημοσιευθούν όλα τα έγγραφα και να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι τι γίνεται. Επί της ουσίας, για δραστηριότητες χωρών όπως η Ισπανία για παράδειγμα, λόγω ανισορροπιών που υπάρχουν μεταξύ των χωρών και των τομέων. Δεν θα αυξηθεί η ζήτηση. Δεν δουλεύουμε λοιπόν γι' αυτό. Υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες λοιπόν να δημιουργηθεί απασχόληση και κυρίως να επαναβιομηχανοποιηθεί η Ευρώπη με ισορροπημένο τρόπο που θα έπρεπε να ήταν μια απόλυτη προτεραιότητα για τη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Έχουμε παραδείγματα άλλων συμφωνιών όπου αυτό γίνεται και ακολουθείται όπως στην ΑΦΤΑ. Ένα εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης που χάθηκαν στα πρώτα χρόνια. Λιμνάζουν οι μισθοί στα επίπεδα πολλών δεκαετιών. Οι Ευρώπη και οι πολίτες χρειάζονται, όπως αναφέρθηκε, οι επενδύσεις στην Ευρώπη. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η απάντηση. Και αυτή η συμφωνία δεν πορεύεται προς αυτήν την κατεύθυνση καθόλου. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Σταλίτσικα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει όντως να ληφθεί υπόψη η γνώμη του Κοινοβουλίου. Δεν ομονοούμε ακόμη, αλλά ακόμα βρισκόμαστε στην διαδρομή. Εγώ πιστεύω στο TTIP και επίσης, όπως και και Αγγέλικα, πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα στην Τσεχία. Πολλές φορές είναι και τεχνητά τα προβλήματα. Θα πρέπει να έχουμε διαφάνεια, αλλά θα πρέπει να είμαστε και συγκεκριμένες τις διαπραγματεύσεις. Δεν λέω όλα να βγουν στη φόρα των διαπραγματεύσεων τα σχετικά. Γι' αυτό είναι σωστό ότι γίνεται σήμερα ενημέρωση. Ας έχουμε ε, περισσότερη ενημέρωση στο μέλλον. Ακόμα και αν γίνεται σε μικρότερο κύκλο η βασική πρόκληση. Επομένως, είναι οι διαπραγματεύσεις αυτέ. Και, πέστε μας κάπως περισσότερα, όσον αφορά τις κρατικές προμήθειε σε σχέση με την ενέργεια. Γιατί είναι αυτό η μεγάλη πρόκληση του τίτλου. Δεύτερον, πυρηνική ασφάλεια. Είναι ζήτημα το οποίο καταρχήν μας έχει διαιρέσει εμάς σε σχέση με τους προελλαντικούς μας εταίρους. Από τη μία μεριά έχουμε ε, την ε, Ρουσία και από την άλλη τους Αμερικανούς. Το, τρίτη, το τρίτο ζήτημα που είναι το πλέον σημαντικό ε, αφορά την τυποποίηση και το ρυθμιστικό περιβάλλον. Θα αντιμετωπίσουμε διοικητικό άχθος με βάση τα όσα συζητούνται και για τις δημόσιες προμήθειες και σε αυτό τον τομέα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, κοιτάξτε, σε γενικέ γραμμέ είμαι υπέρ των ε, ελεύθερων και των ελεύθερων συναλλαγών και των σχετικών συμφωνιών. Αλλά όταν ακούω για το TTIP, ε, πρέπει να καταλάβω κάποια πράγματα για να συμφωνήσω. Μιλάτε για ε, επαναβιομηχανοποίηση, για την στάση του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς τα ίδια ζητούμε. Όμως είναι πραγματικά φαινομενικέ οι διαστάσει που έχει πάρει η συμφωνία αυτή και το πόσο ενδιαφέρει. Τι θα γίνει, α πούμε, με τι εθνικέ υπηρεσίε υγεία, που ε, κάποιε φορέ έχουν, ελέγχονται από το κράτο, αλλά πολλέ φορέ υπάρχει και ιδιωτική χρηματοδότηση. Δεν μιλάω για ε, μια πλάγια ιδιωτικοποίηση αναγκαστικά, αλλά οι ε, πολίτες φοβούνται ότι βάσει αυτής της συμφωνία οι δικηγόροι των ΗΠΑ μπορεί να χρησιμοποιούν το ε, ε, ISDS, δηλαδή το μηχανισμό επίλυση διαφορών από τον επενδυτή προς το κράτος, για να ήσουν λόγω χάρη το κράτο του ΗΠΑ. Βασιλείου. Και πολλέ φορέ ξέρετε ότι οι δικηγόροι που εργάζονται για το Αμερικανικό κράτος είναι δικηγόροι της Νέας Υόρκης. Αυτό λοιπόν μπορεί να σημαίνει ότι στα χέρια σας περνάει και το Εθνικό μα Σύστημα Υγείας. Ευχαριστούμε. Κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ τη συζήτηση θέλω σύντομα για δύο ουσιώδη θέματα να την εμπλουτίσω. Εδώ είμαι, εδώ βρίσκομαι. Ευχαριστώ. Μια και έτσι ξεκινήσατε και πάλι βλέποντας το θέμα της διαφάνειας που από πολλούς συναδέφους δόξα τω Θεώ αναγνωρίζετε και αναφέρετε και εγώ το αναφέρω. Είχατε αρχίσει να λέτε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη λέει διαφάνεια. Η κυρία Επίτροπος στις ακροάσεις δεσμεύθηκε για μεγαλύτερη διαφάνεια. Μια νέα κίνηση λέει θα γίνει σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις TTIP, νέα όθηση, νέα προαγωγή των θεμάτων. Πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά πείτε μας συγκεκριμένα τι έχετε υπόψη σας όταν υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για τη διαφάνεια, ποιες επιλέγετε και τι κάνετε. Ποιες είναι οι 5, 6, 7 δυνατότητες δράσης. Όλοι οι συνάδελφοι που είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο για την TTIP να γίνει κάτι, ο συνάδελφος τα ανέφερε αυτά επί, επί ενός σημείου. Κάνουμε διαφήμιση. Είμαστε υπέρ της TTIP. Πολλές ευκαιρίες θα υπάρξουν σίγουρα. Αλλά πολύ λίγα γνωρίζουμε ακόμη εμείς. Και οι πολίτες έχουν φοβίες, φόβους, ανησυχίες. Υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν την TTIP. Υπάρχει μια εκστρατεία μέσω του διαδικτύου. Δράσεις χωρίς τέλος. Το βράδυ της Δευτέρας ήμουν σε μια τέτοια εκδήλωση. 100 άνθρωποι. Οι 99 είπαν γιατί είναι κατά της TTIP. Και εγώ είπα, δήλωσα, να αναμείνουμε, να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για να κρίνουμε στο τέλος τι γίνεται. Είναι δύσκολο όμως να γίνει αυτό. Ελάτε, ελάτε σε εμά ε, στις εκλογικές περιφέρειες ε, και κάντε εκεί διαφήμιση υπέρ της TTIP. Αν συνεχίσουμε έτσι κυρίες και κύριοι, τότε Μπορώ να προσθέσω τη φωνή μου στην φωνή πολλών συναδέλφων. Μπορούμε να αφήσουμε τα πράγματα να εξελίσσονται ως είναι, αλλά μην εκπλαγείτε στο τέλος όταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακουστεί ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία δεν θα συμπορευτεί προς την κατεύθυνση έγκρισης της TTIP, διότι δεν κατανοούν οι πολίτες και δεν εγκρίνουν όλα αυτά περί των οποίων πρόκειται εδώ. Δεύτερο, Υπάρχουν συγκεκριμένες φοβίες και φόβοι και ανησυχίες των πολιτών. Αυτές και αυτά πρέπει να απαντήσετε με τις τοποθετήσεις σας. Κάθε κοινότητα, κάθε δήμος κάνει εκδηλώσεις κατά της TTIP. Ξεκινώ με τους δικούς μου ψηφοφόρους. Τι γίνεται για να, τους, να πετύχουμε, να τους προσελκύσουμε. Είναι πολύ δύσκολο το έργο μην νομίζετε ότι είναι απλό. Πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα των αρμόδιων για τη δημοτική πολιτική, περιφερειακή πολιτική, κοινοτική πολιτική. Λέγαμε στο Ευρωκοινοβούλιο δεν θέλαμε να έχουμε περαιτέρω φιλελευθεροποίηση και όλα αυτά αποτελούν αντικείμενα διαπραγμάτευση κτλ. κτλ. Πείτε μα λοιπόν τι γίνεται, πρέπει να ολοκληρώσω. Υπάρχουν λοιπόν πολλέ ανησυχίε και ερωτήματα. Αν και στα θέματα ενέργεια έχω και εκεί μια ερώτηση που θέλω να διατυπώσω και για το fracking, για το σχιστολιθικό αέριο τι γίνεται, θα διαπραγματευτούμε και επ' αυτού υπάρχουν ανησυχίε. Υπάρχουν χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θέλουν να προωθεί το fracking, η διάρρηξη, η διαρρογματική εκμετάλλευση ε, του, του αερίου. Όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν λοιπόν. Ο κύριο Παλ Ρούμπεχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ ότι και η Επιτροπή Βιομηχανίας μπορεί να ασχοληθεί και σε βάθος και έντονα με αυτά τα θέματα ενδιαφερόμαστε φυσικά για τις επενδύσεις και τις άμεσες ε, αλλοδαπές επενδύσεις στην Ευρώπη. Ενδιαφερόμαστε οι επιχειρήσεις μας να μπορέσουν να επενδύσουν και στη ΣΥΠΑ. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σαφές ότι η προστασία της ιδιοκτησίας πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο. Στην Ευρώπη αναφέρονται περιπτώσεις όπως εδώ στην Επιτροπή Ενέργειας Δηλαδή η περίπτωση Vattenfall που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με νομολογία του σχετικά. Τι θα γίνει, θα διατηρηθεί χωρίς τη διαδικασία TTIP ή θα είναι ξεχωριστό θέμα στη διαπραγμάτευση με την υφιστάμενη νομοθεσία στην Ευρώπη. Τι θα γίνει. Από την άλλη πλευρά έχουμε και την, ας το πω έτσι, ε, αφαίρεση ιδιοκτησιών ή περιουσίας από τους γεωργούς μας λόγω του ότι μισθώνονται κάποιες ε, εκτάσεις π.χ. στην Ουγγαρία έχουμε πρόβλημα επενδύσεων στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει σχέση με την TTIP αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 10 που θα μπορούσε να αποφασίσει σε περίπτωση ε, επίμαχων θεμάτων. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση με τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρξουν εκεί επίμαχα θέματα. Έχουμε διαδικασίες και ρυθμίσει ρυθμίσει σχετικά. Ποιο θα είναι αρμόδιο για τέτοια επίμαχα θέματα που θα υπάρχει κάποια σύγκρουση. Εδώ δεν θέλουμε εμπορικό πόλεμο, δεν θέλουμε πόλεμο. Θέλουμε να υπάρχουν τακτές και τακτικές διαδικασίες, νόμιμες, με διατάξεις και διαδικασίες, Ποιο θα είναι υπεύθυνο γιατί και να υπάρχει επιδιαιτησία από κάποιο δικαστήριο ή κάποιο φορέα, ιδιαίτερα σημαντικό για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Νομίζω ότι έχει τεράστια σημασία αυτό εμείς έχουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη που εξάγουν. Η μεγάλη ανάπτυξη, η πραγματική ανάπτυξη δυστυχώς διεξάγεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει έναντι της Ευρώπης τα θέματα αυτά απέναντι στη ΣΥΠΑ να τα ενισχύσουμε ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν καλύτερους όρους ε, ανταγωνισμού και επιβίωσης. Είναι σαφές ότι άλλοι αλλού στον κόσμο θα απολέσουν, θα χάσουν. Ξεκινούν εδώ να παρεμβαίνουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως λομπιστές. Βλέπουν που βρίσκονται τα τροτά σημεία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δρούν. Γι' αυτό είναι έργο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ εντονότερα να ενημερώσει. Γι' αυτό ευχαριστώ για το ότι βρίσκεστε εδώ παρόντες εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσετε χειροπιαστές απτές απαντήσεις. Και βλέπετε λοιπόν ότι με αυτή την πορεία πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μπόνη. Το μικρόφωνο σας ξαναπατήστε το, λέει ο κύριος Μπούζεκ. Το TTIP είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, για την ανάπτυξη της Ευρώπης. Θα ήθελα όμως να σας ε, υποδείξω ένα πρόβλημα. Προστασία δεδομένων, ε, καθώς και όροι και προποθέσεις όσον αφορά ε, την οικονομία που αφορά την οικονομική πλευρά τέλο πάντων αυτή τη υπόθεση. Δηλαδή να υπάρχει ανάπτυξη τη οικονομία με την ανάπτυξη αυτών των λεγόμενων big data, των μεγάλων δεδομένων, μεγάλων όγκων δεδομένων, γιατί εμείς περιμένουμε να αποκρισταλώσει η θέση το Συμβούλιο όσον αφορά κάποια δέσμη με τον προστασία των δεδομένων και ε, ε, ε, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει πρώτα πρώτα να ολοκληρωθεί ο σχετικό κανονισμός και να μην αντιπρονατευόμαστε όλα μαζί να, όλα να τα ρίχνουμε στο ίδιο καράθι στα πλαίσια του TTIP. Θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει αυτές οι διαδικασίες να διέπονται από κάποιο συντονισμό. Θα πρέπει να δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, πώς ε, συντονίζει αυτά τα θέματα, πώς εξασφαλίζει την συνέπεια στα δύο μέτωπα και τι κάνει ακριβώς η Επιτροπή ούτως ώστε να κατοχυρώσει τα δικαιώματα των πολιτών σε σχέση με τα δεδομένα. Να δούμε πώς ακριβώς τα πράγματα σχέση με τη συμφωνία Ομπρέλα. Πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά το πώς θα ξεκαθαριστεί ε, αυτή η υπόθεση της προστασίας των δεδομένων. Ο πρόεδρος Μπούζεκ, ευχαριστώ και εσάς γιατί τηρήσατε το χρονικό όρο της παρέμβαση. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή για την ενημέρωση που μας παρήχε και να επισημάνω ότι το ποιο ρόλο θα παίξουν τα εθνικά κοινοβούλια δεν πρόκειται να το αποφασίσουμε εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι υπάρχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω την αρχή των δοτών αρμοδιοτήτων και το τεκμήριο αρμοδιότητες ότι βρίσκεται στα κράτη-μέλη. Από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εδώ πρόκειται σαφέστατα για μια μεικτή συμφωνία, μια mixed agreement που κατά την άποψή μας έχει ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή στο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων τους. Επομένως είναι ξεκάθαρες οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν. Και αν υπάρξει μια υπόνοια ενδεχόμενα περιορισμού των αρμοδιοτήτων των Εθνικών Κοινοβουλίων αυτό θα είναι άσχημο γιατί θα δημιουργήσει υπεραιτέρω αρνητικό κλίμα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν συζητούμε θέματα σε μια διεθνή συμφωνία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, προφανώς εδώ υπάρχουν αρμοδιότητες των κρατών μελών και δεν μπορεί να τις υφαρπάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο θέμα αφορά το τι θα γίνει με αυτή τη μεγάλη συμφωνία, εγώ την ονομάζω το οικονομικό ΝΑΤΟ, Economic NATO αυτή είναι η αντίληψη την οποία βλέπω ότι έχει αυτή η συμφωνία. Θα βοηθήσει τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε ότι οι επενδύσεις επηρεάζονται από τα κόστη και η ανταγωνιστικότητα δεν εξαρτάται μόνο όπως λαθεμένα πιστεύανε αρκετοί από τη μείωση του κόστους εργασίας αλλά κυρίως από το κόστος της ενέργειας. Γι' αυτό και βλέπουμε να εγκαταλείπουν στις ΗΠΑ την αντίληψη του outsourcing και να επιστρέφουν επενδυτές και αμερικανικές εταιρείες εντός των ΗΠΑ, διότι εκεί υπάρχει φτηνή ενέργεια με το σχιστολιθικό αέριο. Επομένως έχω την εκτίμηση ότι δεν θα γίνουν επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντίθετο, επιχειρήσεις μεγάλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επενδύσουν στι Ηνωμένε Πολιτείε αξιοποιώντα το φτηνό σχιστολιθικό αέριο. Άρα θα έχουμε αποβιομηχάνηση σε πρώτη φάση τη Ευρώπη, περιορισμό των επενδύσεων και το αντίστροφο από αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη και να μα ενημερώσετε γι' αυτό, όπω επίση μια κουβέντα μόνο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές, δεν έχουν την εμπειρία να ανταγωνιστούν σε τεράστιες αγορές. Αντίστοιχη εμπειρία έχουν Just a second, Mr. Chairman. Well, Αντίστοιχες εμπειρίες έχουν κυρίω οι επιχειρήσει οι μικρομεσαίες των ΗΠΑ να δουλεύουν σε μεγάλε αγορέ. Πώ θα επηρεάσει αυτό την ανταγωνιστικότητα. Thank you very much. A lot of complaints. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Πολλά παράπονα και δικαιολογημένα, λέει ο πρόεδρο, Αλλά όμω οι προσκεκλημένοι μα τώρα θα επιθυμούσαν να απαντήσουν, αλλά και μετά θα ακολουθήσουν έξι συνάδελφοι για ερωτήσει. Και εδώ σας προτείνω να κλείσει ο κατάλογος των αγορητών γιατί θα πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Συμφωνείτε? Καλώς. Άντε 7. Άντε 7. Καλώς. Τέλος. 7 και κανείς άλλος. Απαντήσατε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν είδη εισαγωγής. Έχω σας πω ότι είμαστε δημόσιοι υπαλλήλοι. Όποτε θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσετε οτιδήποτε. Εάν θέλετε ενημέρωση, Επίσης θα συνεργαστούμε, να έχει γίνει, θα συνεργαστούμε και με τον κύριο Λάγκε στην δική του επιτροπή, αλλά και με τη δική σας επιτροπή πρέπει να συνεργαστούμε. Οποτεδήποτε επομένω έχετε κάποιο ενδιαφέρον, περιέργεια, κάτι να μάθετε, πληροφορίες. Εγώ ή ο Πέτρος θα θα ε, προσφέρουμε όλοι μας την έμπειρο γνωμοσύνη. Πάντως, σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Βουλευτής, όσον αφορά με το ότι θα πρέπει να βγούμε να τα πούμε στον κόσμο με όλο το σεβασμό. Αυτό είναι δική σας δουλειά. Κοιτάξτε, δεν θέλετε να κάνετε τη δική μου δουλειά. Κάθε μέρα κάθομαι στο γραφείο πάρα πολύ βαρετό, μέχρι τις 9 το βράδυ. Οπότε το πώ θα εμπλακούν οι πολίτε, πώ θα του εξηγηθεί περί τίνο πρόκειται και γιατί είναι κάτι το καλό για εκείνου, ποια είναι τα, τα, τα, τα κέρδη από αυτέ τι διαπραγματεύσει, ο πώ ε, τα υπέρ είναι πολύ περισσότερα από τα κατά και από τον ανταγωνισμό από τους ε, Αμερικανούς ε, παραγωγούς. Αυτό είναι θέμα της δημοκρατικής λειτουργίας. Εξαρτάται από εσάς ή από την Επίτροπο. Μία είναι η Επίτροπος, ε, ε είπαμε έχουμε τόσα πολλά κρατημιλια αλλά έχουμε πέντε, πέντε που δουλεύουν για το TTIP. Και ε, υπάρχει βέβαια και εξειδίκευση, άλλο καθένας έχει άλλο θέμα, ε, εξάτομα θα με τι διαπραγματεύσει. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε κάποια όρια. Αλλά τελικά αυτό που μπορεί να γίνει είναι το πώς θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό θέλουμε να αλλάξει. Και κάθε μέρα έλεξε μια ματιά στο, στο ΑΕΠ, το δικό μου και των Αμερικανών και τα δύο μαζί. Πέφτει 45%. Ήμασταν 55% πριν από 10 χρόνια. Πριν από 6 χρόνια ήμασταν στο 65% κάθε χρόνο. επομένω. όλο ένα και πέφτει το ΕΠ, γινόμαστε όλο ένα μειοψηφούντε μέτοχοι κατά κάποιο τρόπο στο παγκόσμιο ΕΠ. Να τι θέλουμε να άρουμε, να αλλάξουμε με την εμπορική πολιτική. Γι' αυτό σας λέω. Μιλούμε για ε, θέμα της Ευρώπης. Κάτι το οποίο φυσικά προποθέτει τη δική σας έγκριση. Για τις ΜΜΕ που ρωτήσατε. Ε, και αυτό είναι και αμερικανική προτεραιότητα. Δεν είναι ότι εμείς θέλουμε τις ΜΜΕ και όχι εκείνη Θέλουμε και οι δύο κάτι να κάνουμε εις αυτήν την υπόθεση που να ωφελεί τις ΜΜΕ. Οπότε, ό,τι προτάσεις έχετε, να μας τις πείτε, διότι αυτή είναι η δουλειά μας. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα εντάξουμε στην συμφωνία. γιατί την προσθέση των δεδομένων τώρα σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Ε, Εμεί προσπαθήσαμε να κάνουμε το διαχωρισμό, γιατί εσείς είπατε ότι προστασία των δεδομένων είναι ευρωπαϊκό δικαίωμα. Κατοχυρώνεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχουμε τον κανονισμό, δεν πρόκειται για ακόμα ένα οικονομικό μέγεθος, ένα οικονομικό δικαίωμα το οποίο επιδέχεται διαπραγμάτευση ή στα πλαίσια της εμπορικής συμφωνίας. Οπότε γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να τα διαχωρίσουμε. Αλλά θα πρέπει να τα ανταποκριθούμε και στο αμερικανικό αίτημα ότι θα πρέπει τα δεδομένα να, να, να υπόκεινται σε κάποια ροή... να υπάρχει τέλο πάντων ανοιχτό ε, πνεύμα στα πλαίσια του TTIP. Αλλά είναι θέμα επομένως και της Ευρώπης και της ε, Αμερικής σε σχέση με την προστασία που θα ορίσουμε. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν σεβαστά από κάποιες εταιρείες οι οποίοι ε, παίρνουν τα δεδομένα και τα βγάζουν από την Ευρώπη και αφορούν τους, τους πολίτες. Και δεν είμαι, δεν είμαι ειδικό σε αυτό, αλλά όσο μπορώ σα τα λέω. Τα για τη διαφάνεια τώρα. Είπαν κάποια μέλη αρκετά. Και... Έκαναν κάποια σχόλια ευρωβουλευτέ ε, και σε σχέση με τι διαπραγματεύσει στι οποίε συμμετείχα εδώ και 25 χρόνια γίνεται αυτή η προσπάθεια. Όλα τα έγγραφα αρχικών θέσεων βρίσκονται στη ιστοσελίδα του διαδικτύου. Όσοι λένε είναι κρυπτό και παραβίστο δεν αληθεύει αυτό, δεν ευσταθεί. 70% των στοιχείων μας είναι στο διαδίκτυο και όλα τα κείμενα που διαπραγματευόμαστε μπορούν να τα συμβουλευτούν τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας και τα, τα κράτη-μέλη τα ίδια. Έχετε λοιπόν πρόσβαση σε όλα και άπαντα επί των θεμάτων που διαπραγματευόμαστε ως κείμενα. Και περνάμε τώρα σε παγιωμένα, ολοκληρωμένα κείμενα με τη ΣΥΠΑ. Και εκεί και πάλι θα είμαστε σε επαφή με τον πρόεδρο Λάνε ώστε εσείς και όχι μόνο τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας αλλά και οι άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα κείμενα. Είναι πολύ στεγνά όμως, ε, δεν είναι τόσο συναρπαστικά. Τίθεται θέματα σωστής κατανόησης του κειμένου, των κειμένων και δουλειά μας είναι να σας διευκολύνουμε να τα κατανοήσετε. Αμφισβητώ οποιονδήποτε λέει και ισχυρίζεται ότι δεν μας ενδιαφέρει η κοινωνία των πολιτών και όλη την ημέρα χθε το απόγευμα το περάσαμε με τον Πέτρο για θέματα κοινωνίας των πολιτών. Δεν ευσταθούν λοιπόν αυτά. Έχουν αναφερθεί στοιχεία και είμαστε βέβαιοι ότι από πλευρά Επιτρόπου Σουηδού που είναι, ενδιαφέρεται απόλυτα για τα θέματα διαφάνειας ότι η ίδια προσέγγιση υιοθετείται. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις προδιαγραφές για τα οχήματα, τα αυτοκίνητα που αναφέρθηκε. Είναι ένα από τα πιο ρυθμισμένα προϊόντα σε παγκόσμια κλίμακα. Αν σκεφτείτε πόσες διατάξεις και ρυθμίσεις πρέπει να είναι σεβαστές και να συμμορφωνόμαστε με αυτές όταν παράγουμε ένα όχημα. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μηχανισμούς ώστε να αναγνωρίζουμε αμοιβαία τις ρυθμίσεις και διατάξεις ε, αμφωτέρωθεν Παράδειγμα, περιβαλλοντικοί κανόνες και κανονισμοί για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τα αυτοκίνητα. Δεν θα είναι απόλυτα οι ίδιοι και ταυτόσιμοι, αλλά προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε τους τομείς εκείνους όπου η αμοιβαία αναγνώριση θα μπορούσε να καταστήσει πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσει μα για την Εθνική Υπηρεσία Υγείας, NHS ε, και το ISDS που αναφέρθηκε πιο πριν. Έχουμε αποσαφηνήσει στην TTIP τα θέματα και είπαμε ότι τα κράτη-μέλη θα είναι, θα είναι ε, ε, ελεύθερα στο μέλλον όχι μόνο να, έχουν, να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες που θα παρέχονται με δημόσια κονδύλια, αλλά επίσης να μπορούν να ε, κρατικοποιηθούν μετά από ιδιωτικοποίηση. Αυτό το πρόβλημα το οποίο ε, βιώνετε εσείς με ιδιωτικοποίηση σε σχέση με την NHS, αν θέλετε να αντιστραφεί αυτό στο μέλλον, θα είναι δυνατό και εφικτό. Θα προστατέψουμε κάτι τέτοιο. Θα βρίσκεται λοιπόν υπό ένα προστατευτικό πλαίσιο. Λοιπόν, ε, το άλλο θέμα που αναφέρεται είναι πάρα πολύ πολιτικού χαρακτήρα και δεν θέλω να εμπλακώ σε κάτι το οποίο θα μπορούσα να πω και να πάει στραβά και δεύτερο, σε αυτό το οποίο ανήκει μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια σε αυτή τη διαβούλευση, το μόνο που θα ήθελα να πω είναι δύο πράγματα. Πρώτον, είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα τώρα. Δεν είναι εθνική αρμοδιότητα πλέον αυτό το θέμα. Ανήκει στα θέματα εμπορίου βάσει τη συνθήκη Λισαβόνα. Αυτή είναι η επιλογή που έκαναν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Δεύτερο, να γνωρίζετε παρακαλώ ότι η ε, διάταξη επίλυση ε, επίμαχων θεμάτων από κράτο σε κράτο δεν προστατεύει πάντα από κράτος σε κράτος ε, τους ε, ε, επενδυτές. Είναι θέματα εμπορίου που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υπό μη διακριτική μεταχείριση. Δεν λειτουργεί όμως αν έχετε μια μικρή επιχείρηση που οι επενδύσεις της για παράδειγμα δημεύθηκαν ή κατασχέθηκαν. Αυτό που προσπαθούμε να εντοπίσουμε και να ταυτοποιήσουμε είναι ένα σύστημα που θα σέβεται τις δημοκρατικές αρχές. Ταυτόχρονα όμως θα σέβεται και αυτές τις αρχές διότι στην Ευρώπη Ευρώπη είμαστε μια ε, οικονομία που βασίζεται στη γνώση και έντονη εκμετάλλευση κεφαλαίου, κεφαλαιοκρατικής χρήση. Σας ευχαριστώ. Εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Για θέματα ενέργειας τώρα και για το θέμα το οποίο τίθεται για το γεγονός ότι δεν έχουμε μια κοινή αγορά ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς αυτό επηρεάζει τις διαπραγματεύσεις. Όπως γνωρίζετε, μία από τις κύριες προτεραιότητες ε, της Επιτροπής Juncker είναι ακριβώς το να κινηθούμε και να προχωρήσουμε προς μια ενεργειακή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό αντανακλάται επίσης με τον τρόπο που αυτοδιοργανώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αντιπροέδρους, ε, με αρμόδιους για ε, τα συναφή θέματα. Αντιλαμβανόμαστε φυσικά ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να επιτευχθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να επιτευχθεί η Ενεργειακή Ένωση. Δεν θα γίνει μια νυχτή μέσω κάποιων απλών διαπραγματεύσεων. Όμω οι διαπραγματεύσει TTIP μπορούν να συνεισφέρουν και να συνδράμουν ώστε να επιτευχθεί αυτό ο στόχο. Και διτά αυτό. Πρώτον, αναφερόμενος σε μία από τις σημαντικές διεκδικήσεις μας, δηλαδή την άρση των εξαγωγικών περιορισμών όσον αφορά προϊόντα όπως το φυσικό αέριο και το ακαθάριστο αργό πετρέλαιο. Αυτό φυσικά αναγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε την πρόσβαση που θα είχαμε στις διεθνείς αγοράς ενέργειας. Πρώτον, θα διευκολύνει την αποκερμα κερματικοποίηση αγορών σε σχέση με τα προϊόντα αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια αυθεντική παγκόσμια αγορά και καθώς ε, οι ε, διάφορες, διάφοροι περιορισμοί πρέπει να αντιμετωπιστούν για να μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε προς μια πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά σε αυτό το επίπεδο που μπορεί να μας ε, βοηθήσει ώστε να επιτύχουμε μειωμένες τιμές, μειούμενες τιμές και την διαφορά τιμών που ένα, ένας άλλος ευρωβουλευτής ανέφερε συγκεκριμένα όταν είπε ότι για παράδειγμα λόγω των ενεργειακών τιμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαμε να κινητοποιηθούμε, να κινηθούμε προς μια πιο παγκοσμιοποιημένη αγορά που θα βοηθούσε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μειώσουν τις ε, τιμές, τη διαφορά τιμών για τα ενεργειακά προϊόντα που τις ε, ε, αφήνει πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ και τον μεγάλο προσανατολάς εταίρο μας που είναι ο κύριος πάροχος ενεργειακών προϊόντων, ιδιαίτερα φυσικού αερίου, δηλαδή τη Ρωσία και να υπάρξει απεμπλοκή και να έχουμε μια πολυμορφία, πολυμορφοποίηση των δυνατοτήτων ανεφοδιασμού μας με ενεργειακά προϊόντα. Κάτι τέτοιο θα ήταν μια σημαντική συνεισφορά. Μια συγκεκριμένη λοιπόν συνεισφορά. Το δεύτερο αφορά τη δημιουργία εν μιας δυνατότητας να υπάρξουν κανόνες και κανονισμοί που θα είναι σεβαστοί στο μέλλον και θα προσαρμόζονται προς αυτούς τρίτες χώρες. Εφόσον θα συμφωνούσαμε με αυτούς σε αυτούς τους κανονισμούς με τη ΣΥΠΑ θα μπορούσαμε αντί τρίτων χωρών να προτείνουμε τους ίδιους κανόνες και κανονισμούς αυτοί να γίνουν δεκτοί και από τρίτα κράτη και να κινηθούμε σταδιακά προς παγκοσμιοποιημένους κανόνες και πλαίσια διατάξεων που θα είναι ενιαία. Αυτό μια και σήμερα σε σχέση με τις τρίτες χώρες δεν θα αλλάξει ξαφνικά το πλαίσιο άμεσα είτε και ε, ε, μεσοπρόθεσμα. Είναι μακροπρόθεσμο αυτό το εγχείρημα. Υπήρξε και μία ερώτηση για τις δημόσιες προμήθειες ε, όσον αφορά ενεργειακά προϊόντα. Αυτό πρέπει να ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση και διαπραγματεύσεις για τις δημόσιες προμήθειες. Όπως θα έχετε κατανοήσει, είναι ένα πεδίο αυτό για την διεξαγωγή μιας επιθετικότερης, επιθετικότερης πολιτικής υπέρ των ευρωπαϊκών συμφερόντων που δεν στέφθηκε ακόμα με επιτυχία αλλά θα πρέπει και να συζητηθεί και να συνεχίσει στο μέλλον. Και θέματα πυρηνικής ασφάλειας. Θέματα πυρηνικής ασφάλειας δεν ρυθμίζονται μέσω αυτής ειδικά της συμφωνίας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη συμφωνία μεταξύ Ευρατόμ και των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα πυρηνικής ασφάλειας και ενέργειας. Και το τελευταίο που ανέφερε η κυρία Νίμπλερ, για την διαρρογματική εκμετάλλευση συστολιθικού αερίου. Και πρέπει να πω ότι εδώ τίποτα σε αυτή τη συμφωνία δεν θα έχει επιπτώσει στα κυρίαρχα δικαιώματα κάθε συμβαλόμενου μέρους για τις αποφάσεις που θα λαμβάνει για την εκμετάλλευση φυσικών του πόρων. Και όταν λέω συμβαλόμενα μέρη, φυσικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό σημαίνει τα κράτη-μέλη. Για τη ΣΥΠΑ σημαίνει τις επιμέρους πολιτείες πολιτιακά. Για την, ε, το συστολιθικό αέριο στη ΗΠΑ υπάρχουν κάποιε πολιτείες που αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα του συστολιθικού αερίου. Και κάποιες άλλες πολιτείες που αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση, να μην επιτρέψουν τέτοια εκμετάλλευση του συστολιθικού αερίου. Η ίδια κατάσταση υπάρχει ακριβώς και σε ΣΥΠΑ. Υπάρχουν άλλα κράτη-μέλη που είναι περισσότερο υπέρ, άλλα κράτη που δεν θέλουν να εμπλακούν σε αυτή την προσπάθεια και τίποτα σε αυτή τη συμφωνία δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα κράτη-μέλη μας και να μπορούν να λαμβάνουν κυρίαρχα αποφάσεις επ' αυτού. Ευχαριστώ. Έχουμε 7 ερωτήσεις. Ένα λεπτό ένα ερώτηση. Κύριε Στανίσου. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Η ερώτησή μου πάλι αφορά την επικοινωνιακή μας πολιτική. Πιστεύω στι καλέ σα προθέσει να είναι διαφανή οι διπλωματεύσει, όμω έχει ριζώσει βαθιά η καχυποψία ότι η συμφωνία TTIP θα χρησιμοποιηθεί για να αλλάξει όλο το κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαφέρει αρκετά των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να γνωρίζετε από αυτή την πλευρά ε, οι οικονομικές ε, ερωτή, παράμετροι έχουν δεύτερη, έρχονται δεύτερες όταν η κοινωνία είναι τόσο ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα. Άρα είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια πολύ ενεργό επικοινωνική πολιτική. Εφόσον η ουσία είναι καλή, ε, περάστε στην ουσία. Ιδάλλως, το κοινοβούλιο μας, ε, είχατε καμία αρνητική εμπειρία με την άκτα, εφόσον όλα παρουσιάζονται ωραία, φαίνονται καλά, αλλά οι κοινωνίε δεν συμφωνούν, δεν είναι ενημερωμένε, υπάρχουν υποψίες ότι οι θεμελιώδει ελευθερίε και τα δικαιώματά του θα παραβιαστούν, ε, στο τέλο θα διαμαρτυρηθούν και το κοινοβούλιο θα καταψηφίσει. Αφορά και τη δική σας επικοινωνική στρατηγική. Ε, να επικεντρωθείτε και να μιλάτε παντού. Ευχαριστούμε ο κύριος Βιντάλ. Ευχαριστώ πολύ. Συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτή η διαδικασία της ολοκλήρωσης για το TTP θα περιλάβει ή θα περιλάβει μέσω πρόθεσμα την συγκρότηση κάποιων ε, ε, συμπράξεων ε, ιδιωτικού δημοσίου τομέα γιατί αυτό είναι κλειδί ούτως ώστε να πετύχουμε όπως η μεγάλη τεχνολογική Αμερικανή όμιλη και επίσης νομίζω ότι πρέπει να καταδικάσουμε κάποιο είδους προκαταλήψεις που, που, ανεδίθησαν σήμερα εδώ στην αίθουσα, ότι δηλαδή η τεχνολογία είναι δυνατόν να περιοριστεί, να αλυσοδεθεί, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ και ότι ε, όποιος ε, έχει το, προβάδισμα στην τεχνολογία ε, δεν έχει πάρει σπίτι του και θα είναι για πάντα πρωτοπόρος, επίσης ο προστατευτισμός και αυτό είναι τραγικό και επίσης δεν θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδους αιμονή αντιαμερικανισμού, το καταδικάζω. Ευχαριστούμε κύριο Ζωρίνιο. Ευχαριστώ. Επί της αρχής είμαι υπέρ της συμφωνίας TTIP. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία για να πετύχουμε να ε, εξορροπήσουμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες μεταξύ Ατλαντικού και να φτάσουμε και στον Ελληνικό. Ε, μεταξύ των δύο χθών του Ατλαντικού δηλαδή και να φτάσουμε και στην άλλη του όμως, για όσους ε, έχουν εδώ κάθε λόγο να βρίσκονται στην ε, αίθουσα και να ακούν τη συζήτηση, είμαστε κατά. Δεν είναι περίεργο αυτό. Ε, έχουμε, δεν έχουμε καθόλου παραδείγματα, ή μάλλον έχουμε μόνο αφηρημένα στοιχεία και καθόλου συγκεκριμένα. Να σας δώσω εγώ ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτή την εβδομάδα στην Πορτογαλία υποβλήθηκε έτοιμα στο Δημοτικό Δικαστήριο για να γίνεται η επίλυση των διαφορών με διατησία. Η διατησία, ε, όμως όπως γνωρίζουμε, ε, εξυπηρετεί τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και η πορτογαλική δικαιοσύνη είπε ότι είναι νέας γενιάς απόδοση δικαιοσύνης η διατησία. Αυτά είναι ωραία λόγια. Εάν ε, ένα κράτος θέλει να κρατικοποιήσει ε, το σύστημα υγείας του, μπορεί. Αλλά οι Αμερικανοί μπορούν να διαγωνιστούν και να μπλοκάρουν την όλη διαδικασία το ίδιο και για την υδροοργμάτωση. Ευχαριστούμε συνάδελφε, ο Πρόεδρος. Επόμενος ο μιλητής, ο κύριος Χάνκελ. Δική μου σειρά είναι λέει ο κύριο Χέσκελ, Χέγκελ, συγγνώμη. Ε, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω 100% με αυτό το αίτημα, ότι δηλαδή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι να κάνει παραπάνω για να βελτιώσει την επικοινωνία. Και ο υποφαινόμενο επίση συμφωνεί. Δεν έχω καμία, κανένα δισταγμό να υποστηρίξω αυτή τη συμφωνία με τα στοιχεία που έχω σήμερα. Από την άλλη μεριά, οι περισσότεροι από του. 750 βουλευτές εδώ πέρα δεν ξέρω αν θα συμφωνούσαν γιατί είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα και δίνουμε μια μάχη κατά ενός στρατού εκείνων που δεν αγαπούν την επιχείρηση, την παγκοσμιοποίηση, δεν αγαπούν την Αμερική. Εγώ τα βλέπω καθαρά επαγγελματικά τα πράγματα και πρόταση μου είναι κύριε Πρόεδρε ε, ε, να προτείνει η Επιτροπή μας προς τον κύριο Γιούγκερ, γιατί είχε πει ο Γιούγκερ ότι πρόκειται για κορυφαία προτεραιότητα, μία από τι δέκα κορυφαίε μα προτεραιότητε, να συγκροτήσει ένα γραφείο επικοινωνία. Ε, εκεί να έχουν πρόσβαση όλοι οι βουλευτέ, ε, οι ευρωβουλευτέ τέλο πάντων. Και ό,τι θέμα, ό,τι, ό,τι ερώτηση, απορία έχουν να τη στέλνουν σε αυτό το γραφείο και σε 10 λεπτά να τους απαντούν, τόσο ώστε να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία. Γκρίφιν. Γκρίφιν. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ε, περάσει το μήνυμα το ότι στη, τι πρεσβεύει το νομένο Βασίλειο για το TTIP. Νομίζω ότι μας ε, διασκεδάσατε τις ανησυχίες, αλλά πέστε μας τι συγκεκριμένο κάνετε, ούτως ώστε να εξαφαλίσετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα θέσει σκίνδυνο το εθνικό μας σύστημα υγείας και ε, της ε, κοινοφιλής δημόσιας υπηρεσίας. Δεν θα γίνει τίποτα τέτοιο σήμερα ή αύριο. Επίση, τη μέτρα αναβάνεται ούτω ώστε η κυριαρχία των εθνικών κυβερνήσεων δεν πρόκειται να ψαλιδιστεί και συγκεκριμένα ε, με το ISDS. η κοινωνία το ζητεί αυτό, να διαδυσυχάσετε. Τα συνδικάτα. Ε, και θα πρέπει αυτό να πείτε ιδίως αυτή την υπόθεση το, για τους, για τους επενδυτές, την ε, συμφωνία για τις επενδύσεις ISDS. Ο επόμενος. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να δούμε ότι όλες οι μελέτες για την Αυστρία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, όλες οι μελέτες καταδεικνύουν ότι θα ήταν ένα προτέρημα αμφωτέρωθεν αν υπογράφαμε και οι δύο πλευρές αυτή τη συμφωνία. Οι μελέτες σε σχέση με τη ΣΥΠΑ λένε και δείχνουν ότι μέχρι 750.000 250.000 νέες θέσεις απασχόλησης θα δημιουργηθούν, λέει. Νέες θέσεις απασχόλησης. Ακόμα και σε εμά ε, το κέρδος θα ήταν περίπου 160 δις όλο, όλη η Ευρώπη και παγκόσμια κατά 28% θα σημειώνει αύξηση. Αυτές τις πληροφορίες πρέπει να τις παρουσιάσουμε, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πιστούν. Αν δεν το πούμε με σαφήνεια αυτό, θα έχουμε προβλήματα. Με, μιλώντας για τις λεπτομέρειες, μπορεί ίσως να είμαστε επιτυχείς. Αυτό όμως δεν επαρκεί. Πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες. Ευχαριστώ. Επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία τελικά είναι το μήνυμα. Ε, ίσως και τεχνολογία. Κάποτε μου είπαν ότι στι εμπορικέ διαπραγματεύσεις το πώς αντιλαμβάνεται κανείς τα πράγματα είναι και η πραγματικότητα. Αυτό ισχύει και για εδώ. Η αντίληψή μας ε, καθορίζει την πραγματικότητα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, ότι υπάρχουν θέματα που θα έπρεπε να τύχουν κάποιε μεταχείρισει συγκεκριμένε, αλλά είμαστε πολύ μικρή ομάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπολογίζουμε πάρα πολύ σε εσά και σε όσου μπορούν να πολλαπλασιάσουν το θετικό αντίκτυπο τη ε, επικοινωνία. Κάποιοι θα μπορούσαν να καλύψουν από το χάσμα, είτε είναι υπέρ είτε κατά τη διαφάνεια, ε, γιατί αυτό κάνει μια εμπορική συμφωνία. Ουσιαστικά απελευθερώνει τι αγορέ, είτε το θέλετε είτε όχι. Οπότε ο καλύτερος τρόπος είναι να γίνει με γνώση των στοιχείων και των λεπτομεριών. Προσπαθούμε να δώσουμε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορούμε στον ιστοτοπό της DigiTrade. Σας καλώ λοιπόν να πάτε στη σελίδα αυτή και να δείτε τα έγγραφά μας που είναι δημόσια για να βελτιώσετε τις γνώσεις σας. Ε, είδα προτάσεις προς την Επιτροπή μας, προς τον Επιτροπό μας να βελτιωθεί η σελίδα αυτή γιατί ο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν πρόκειται να επηρεαστούν. Δεν νομίζω ότι μπορώ να είμαι πιο σαφής. Έχει επιβεβαιωθεί και από τους Αμερικανούς. Θέλουν ακριβώς το ίδιο για το δικό τους ε, σύστημα υγείας και για τις υπηρεσίες που παρέχονται υπό την αιγίδα της Αμερικανικής κυβέρνησης. Έτσι το ορίζουν οι Αμερικανοί, οι Αμερικανοί στην νομοθεσία τους. Οπότε αυτό πρέπει να το εγγράψουμε, διότι τα κράτη-μέλη θα είναι ελεύθερα να απελευθερώσουν, να πειραματιστούν με τις αγορές και την παροχή υπηρεσιών στις αγορές, εάν θέλουν να είναι κρατικές υπηρεσίες τους μπορούν να το κάνουν. Για το ISDS, την, το Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών Επενδυτών Κράτους, ε, εδώ το εργαλείο αυτό δεν μπορεί να ε, αμφισβητήσει το δικαίωμα της κάθε κυβέρνηση να ρυθμίζει τα πράγματα, να νομοθετεί. Το μόνο που επιτρέπει αυτή αυτό το εργαλείο, αυτός ο μηχανισμός, είναι να παρακολουθεί τις ζημιές που τις κοιτάζουν οι υπεύθυνοι τη διαιτησία. Δεν κοιτάει όμω ε, η διαιτησία εάν η νομοθεσία ισχύει ή όχι. Δεν επιτρέπεται να το κάνει αυτό. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι λόγω χάρη για την υπόθεση Βάντρεμπελ στην ε, Γερμανία. Η Βάντρεμπελ διαπραγματεύεται με τη γερμανική κυβέρνηση, υπάρχει μια αντίδραση. Οι Γερμανοί αποφασίζουν σταδιακά να καταργήσουν την πυρηνική ενέργεια. Έχουν το δικαίωμα, αλλά μετά αν θέλουν μπορούν να δώσουν αποζημιώσει μα εξαρτώνται από την σύμβαση κύριε και κύριοι. Εάν έχετε τέτοια σύμβαση θα μπορούσε κανείς να απολύσει πυρηνική ενέργεια στη Γερμανία για τα επόμενα 30 χρόνια και κάποια στιγμή ε, να πληρωθεί και μια αποζημίωση εφόσον η κυβέρνηση χάνει στην ε, όλη ε, διαπραγμάτευση. οι Αμερικανοί έχουν χάσει ήδη μια υπόθεση μόνο στο ISDS ως κυβέρνηση. Είναι σπανιότατο. Είναι λοιπόν μια μόδα αυτό που έχει κυκλοφορήσει, μια φήμη. Μερικά θέματα που παίρνουν μεγάλες εκτάσεις σε επίπεδο κοινωνίας είναι πολύ απλό να τα απαντήσουμε. Να πούμε ότι δεν εμποδίζει τις εθνικές κυβερνήσεις ένα τέτοιο ζήτημα να, ε, να νομοθετούν, ούτε επηρεάζει τα δικαιώματα των πολιτών. Ε, ε, μια, ένα σώμα διατησίας κοιτάζει μόνο κατά πόσον υπήρξαν ζημιά και ποιος είναι υπεύθυνο, όχι αν ισχύει η νομοθεσία ή όχι. Τώρα φαίνεται να έχει γίνει μια διευρυμένη συζήτηση αυτή για τις κρατικές πολιτικές. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά εμεί ω επίσημοι υπάλληλοι πρέπει να σα δώσουμε τι ε, ε γνώσει που έχουμε για να σα ε, νομιμοποιούμε στο ρόλο σα. Όταν πάτε σε μια τηλεόραση, σε ένα κανάλι, εσεί ε, νομιμοποιήστε να είστε εκεί. Εμεί όχι. Είμαστε απλώ υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εσεί να εξηγήσετε τι σημαίνουν όλα αυτά, εσεί να του ε, δώσετε να καταλάβουν την ουσία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να είμαστε όσο πιο διαφανεί μπορούμε καταλαβαίνουμε ότι η αντίληψη των πραγμάτων πρέπει να αλλάξει. Η συμφωνία αυτή είναι τόσο μεγάλη που όλοι θα έχουν κάτι να πούνε σχετικά. Και το λέω με κάθε ταπεινοφροσύνη ω ε, δημόσιο υπάλληλο μπροστά σε εκλεγμένου, ερετού ε, πολιτικού ευθύνοντε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Όπω βλέπετε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική συζήτηση για του περισσότερου από εμά. Και Παρ' όλα αυτά, τέθηκαν και συγκεκριμένε ερωτήσει για την ενέργεια, τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Οι συνάδελφοι από την Επιτροπή ΙΝΤΑ ε, επίσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να έχουν όλο και τα περισσότερες πληροφορίες. Γι' αυτό ξαναδίνω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής ΙΝΤΑ, τον κ. Μπεν Ναι, πράγματι. Και νομίζω επίσης, πρόεδρε Μπούζεκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα όσον αφορά τη διαφάνεια και την επικοινωνία. Διότι συχνά το ζω, το βιώνω, ότι πολλές φορές αντικειμενικά μιλάμε για την TTIP, αλλά στο τέλος τέλος ναι. ακούγεται η πρόταση «Δεν εμπιστεύομαι όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Ας προβληματιστούμε να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, κλίμα εμπιστοσύνης και να προωθήσουμε την εμπιστοσύνη και να την κερδίσουμε. Τα ουσιοδέστερα έγγραφα πρέπει να δημοσιοποιούνται πιστεύω. Και για τον τομέα υγείας παράδειγμα. Γιατί η προσφορά όσον αφορά τις υπηρεσίες που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δημοσιοποιείται. Είναι σαφές. 150 τομείς εξαιρούνται. Ιδιαίτερα ο τομέας υγείας, για παράδειγμα. Κάτι τέτοιο θα αντικειμενοποιούσε, θα διευκόλυνε πολύ με αντικειμενικά στοιχεία τη συζήτηση. Αυτή την πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε. Σαφών διατάξεων και σαφών αντικειμενικών τοποθετήσεων. Φυσικά υπάρχει, υπάρχουν κριτικά σημεία, όπω αφορά το ISDS για παράδειγμα. Με κριτικό πνεύμα πρέπει να προσεγγίσουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε διαβουλεύσει ε, όσον αφορά το ISDS ε, και θα καταλήξουμε στο τέλο πώ θα κρίνουμε και ποια συνέχεια θα δώσουμε στις διαπραγματεύσεις επ' αυτού. Λοιπόν, ή δυνατόν διαφάνεια στις συζητήσεις ώστε να, μπορεί, να μπορούν όλοι μας να έχουν αυτές τις πληροφορίες, αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή τους. Και πιστεύω ότι ήρθε πια η χρονική στιγμή επιτέλους η συζήτηση να ολοκληρωθεί με έναν απολογισμό, με μια αξιολόγηση που θα κάνουμε. Επί 1,5 χρόνο, 1,5 έτη συζητούμε με τις ΗΠΑ. Έχει αποσαφινιστεί ποια οδός ακολουθείται, πώς θα πορευτούμε, μπορούμε να συνεννοηθούμε επ' αυτού και περισσότερο για τα χημικά ίσως όχι, αλλά για τα άλλα θέματα. Στον τομέα των δημόσιων προμηθειών και όσον αφορά τέτοια θέματα επί των οποίων είναι εφικτό να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με κριτικό πνεύμα να κάνουμε ένα απολογισμό και να δούμε ποια συνέχεια θα δώσουμε. Αφενός έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφετέρου έχουμε από χθε κιόλα ένα νέο κογκρέσο και μια νέα γερουσία στη ΣΥΠΑ. Και θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό σήμερα η λήψη απόφασης για να γίνει ένα ψήφισμα που θα κατατεθεί για ένα ενδιάμεσο απολογισμό, μια ενδιάμεση αξιολόγηση, το έκανα αυτό, την παρουσίασα αυτή την πρόταση. Μια πρόταση τέτοια να γίνει. Όλες οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν και η Επιτροπή Ήτρε. Και μετά Φεβρουάριο-Μάρτιο θα κάνουμε μια τελική αξιολόγηση. Πού βρισκόμαστε τελικά. Και θα δώσουμε την επισήμαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια συνέχεια θα πρέπει να δώσει στις διαπραγματεύσεις αυτές. Ευχαριστώ. Uh, uh, Ευχαριστούμε συνάδελφοι για προς Τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε και Ίντε προς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διάλογο θα είναι στις αρχές της επόμενης χρονιάς, μετά τον ολοκληρωτό 8ο γύρο διαπραγματεύσεων, σχεδόν αμέσως μετά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ε, όπως γνωρίζετε, η παρουσία σας είναι άκρος απαραίτητη. Ενδιαφέρει τους ίδιους τους πολίτες μας το θέμα. Σας ευχαριστώ. Okay. Ε, Ωραία. Συνάδελφοι, επόμενο σημείο στην ημερήσια διαταξή, εξίσου σημαντικό. Άσερ. Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. Ε, τρίτο πακέτο δεσμημέτρων για την ενέργεια. Γεια σας. Με συγχωρείτε, μην πάτε από εκεί, είναι κλειστά. Μονόδρομος. Ε, ε, Έκθεση για παρακολούθηση της αγοράς και άλλες δραστηριότητες. Η παρουσίαση θα γίνει από τον Αλμπέρτο Ποτότσνικ, τον διευθυντή της Άσερ και τον Λόρδο Μόγκ, πρόεδρο του Συμβουλίου Ρυθμιστών της Άσερ φυσικά. Thank Um, Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια. Η Επιτροπή Ήτρε έχει επιβεβαιώσει και έχει αναθέσει στην αρμόδια ομάδα τη, έχει μάλλον ε, αναθέσει στην αρμόδια ομάδα της για τα θέματα της ΆΣΕΡ να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του οργανισμού αυτού και να συναντιόμαστε συστηματικά με τους εκπροσώπους σας σε διαφορετικά επίπεδα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό ακόμη και σε εθνικό επίπεδο. Και εκεί πρέπει να συναντούμε τους ρυθμιστές μας για να βλέπουμε τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Είναι και ευθύνη μας. Η έκθεση παρακολούθησης της αγοράς είναι πολύ σημαντική, διότι αποτελεί τη βάση για την υπόλοιπη νομοθεσία μας, το τρίτο πακέτο για την ενέργεια, χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει η εσωτερική αγορά ενέργειας, για να γίνει πραγματικά λειτουργική. Ε, πρέπει λοιπόν να ε, σκεφτούμε ότι τα κάτι μέλη δεν πρέπει να αποφασίζουν μόνα τους. Έχουμε στα χέρια μας όλους τους κανόνες, το σύνολο των κανόνων. Αλλά τι θα γίνει με τις λεπτομέρειες με συγκεκριμένα σημεία. Εσείς εκπροσωπείτε ε, και έχετε αναλάβει το δυσκολότερο κομμάτι της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς. Δηλαδή τα κράτη-μέλη πρέπει να μποροντήσουν πλέον να γίνουν δυνατές οι συναλλαγές ενέργειας. Κύριε Ποτότσνικ. Αγαπητοί Ευχαριστώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, ο Ποτότσνικ, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι διότι μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τη δραστηριότητα της υπηρεσίας μας σε σχέση με το έργο μας λοιπόν είχαμε παρόμοια ευκαιρία και στο παρελθόν και επομένως ξέρουμε ότι πάντα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον. Πρέπει είναι και για σας χρήσιμο επίσης μας ε, τιμά η επιλογή σας και το ότι το Κοινοβούλιο ανέκαθεν έχετε δώσει στην ε, ε, η υπηρεσία μας από τότε που συγκροτήθηκε αυτή την ευκαιρία και ιδίω η Επιτροπή Ήτρε. Και ε, είναι επομένω μια πάρα πολύ ε, θετική η εμπειρία που έχουμε με την ομάδα επαφής Acer και έγιναν δύο επισκέψεις αντιπροσωπιών τον Αύγουστο του 2012 και πιο πρόσφατα φέτος. Η υπηρεσία μας συγκροτήθηκε στα πλαίσια του τρίτου πακέτου για την ενεργειακή πολιτική. Για να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές και πρόκειται για θεσμικό όργανο, ευρωπαϊκό, υπόλογο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπαθούμε να προωθήσουμε την ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς, την εναρμόνιση των πλαισίων, των κανονιστικών και επίσης την ακυρότητα της αγοράς σε σχέση με τους στόχους της ελληνικής πολιτικής μας, ούτως ώστε να υπάρχει όφελος εξ αυτού για τους α, καταναλωτές. Ακριβώς συντονίζοντας τις εθνικές αντίστοιχες αρχές. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι το να θίξουμε πέντε διαφορετικές θεματικές ενότητες σύντομα, τόσο ώστε στη συνέχεια να έχουμε αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις σας. Πρώτα, πρώτα, αυτή την έκθεση για την ε, εποπτεία, την θεώρηση της αγοράς. Ε, περσμένη μήνα αφορά το Acer και τις προσπάθειες που έχουν γίνει και Αυτά υπάρχουν στην ε, ιστοσελίδα μας. Είναι μεγάλο αυτό το εργαλείο, πάνω από 25 σελίδες, πολλές πληροφορίες εκεί. Οπότε τώρα απλώς θα δούμε συγκεκριμένα σημεία αυτές της έκθεσης. Επίσης να δούμε ε, πού βρισκόμαστε όσον αφορά την ολοκλήρωση της ε, εσωτερικής αγοράς ενεργείας που είναι ο στόχος του 2014 όπως λέμε. Στη συνέχεια δε μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τα βασικά θέματα του προγράμματος εργασιών μας κατόπιν την πρωτοβουλία που ονομάζεται Γέφυρα προς το 2025. Και επίσης θα δούμε τι γίνεται όσον αφορά την εφαρμογή του σχετικού κανονισμού για την ενέργεια και την διαφάνεια αυτή η αγορά εποπτείας, η, η, η έκθεση ε, θεώρηση της αγοράς αφορά πρώτα πρώτα τις αγορές ε, ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Αφορά τις ε, χονδρικές πωλήσει ε, αυτών των μορφών ενεργείας. Και τα βασικά στοιχεία, το βασικό στοιχείο το οποίο αναδύεται από αυτή την ανάλυση μας στην έκθεση είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει ε, περίπου και πέρσι, ότι δηλαδή οι τιμές λιανικής συνεχίζουν να αυξάνουν παρά το ότι βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα η ζήτηση στα περισσότερα κράτη-μέλη για τον ηλεκτρισμό που μειώθηκε το 2013 ως ζήτηση εις 19 κρατημέλη και η ζήτηση για το φυσικό αέριο το 2013 μειώθηκε σε 17 κρατημέλη. Αλλά αυτό δεν είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές λιανικής. Τα νοικοκυριά πλήρωσαν περισσότερα σε 25 κρατημέλη και στην Ορβηγία εκτός από την Ουγγαρία. Ε, επίσης, άλλο αποτέλεσμα της ε, ε, ανάλυσης είναι ότι σε κάποια κρατημέλη οι φόροι, οι χρεώσεις, τα τέλη καθορίζουν τις τιμές της λιανικής και τις έχουν αυξήσει. Οπότε έτσι έχουμε συρρήγνωση της μεταβλητής ενέργεια ως εμπόρευμα σε λιγότερο από το 50% των ε, τιμών για τον τελικό καταναλωτή. Και δεν μπορούμε να δούμε να υπάρχει κάποιο σχετισμό μεταξύ των τιμών χονδρικής και του ενεργειακού στοιχείου για ε, τις ε, τιμέ λιανικής σε κάποια κράτη-μέλη. Άρα, εδώ πέρα τα πράγματα λειτουργούν όπως θα θέλαμε. Επίσης, έχουμε διαπιστώσει ότι τα νοικοκυριά διστάζουν να αλλάξουν πάρα 6% είναι κατά μέσο όρο το ποσοστό αυτών που έχουν αλλάξει πάροχο. Κάποιες από τις αιτίες του φαινομένου ή έχουμε δει ότι είναι το ότι δεν υπάρχει ενημέρωση, ότι οι τιμές ε, είναι νομοθετικά ε, καθοριζόμενες ε, επίσης ε, η, η πίστη προς τους ε, νέους εργόμενους στην αγορά αλλά και το ότι θεωρούν οι άνθρωποι ότι είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία της αλλαγής παρόχου. Επίσης διαπιστώθηκε ότι σε κάποιες αγορές, κάποια κρατημέλη, και λειτουργεί καλά το σύστημα, σε Βέλγιο, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και κάτω χώρε και στην Νορβηγία για τον πληθυσμό. Γιατί εκεί είδαμε ότι εκεί πέρα είναι περισσότερο ποσοστό αυτών που αλλάζουν πάροχα από ό,τι στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Επομένω, βασικό ε, συμπέρασμα όσον αφορά αυτή την ε, λιανική πόλη ότι θα πρέπει να βελτιωθεί ο ανταγωνισμό σε αυτή την λιανική αγορά. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλαμε, δεν έχουμε μια ανταγωνιστική αγορά. Ακόμα υπάρχουν κάποιοι φραγμοί εισόδου σε αυτή την αγορά και πάντω ε, τα περισσότερα κρατημέλη έχουν περιχαρακώσει το τι ισχύει σε σχέση για τους καταναλωτές, αλλά η προστασία τους ε, έχει ποικιλία μέσων και υπάρχουν πάρα πολλές ε, διατάξεις στον νόμο για την προστασία των καταναλωτών που εφαρμόζονται. Αλλά θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο. Επομένως, η δική μας σύσταση είναι ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την άρση των φραγμών, ούτως ώστε να βελτιωθεί ο ανταγωνισμός. Και επίσης να δούμε πώς θα σταματήσουν να ρυθμίζονται νομοθετικά οι τιμές και επίσης χρειάζεται η εφαρμογή μέτρων των καταναλωτών. Τώρα, πάμε στην πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση της ενεργής αγορά ενέργεια. Και εδώ πέρα ξεκινούμε. Αυτής εξ αρχής, από τότε που ανέλαβε η υπηρεσία μας αυτό το έργο του συντονισμού ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε μια παράλληλη διαδικασία, ώστε να μπορέσουμε να ωφελήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τους ε, καταναλωτές. Οπότε πέραν της, ε, των επισήμων κατευθυντηρίων γραμμών έχουμε και κάποια ε, άτυπη προσέγγιση εφαρμογής για να μπορέσουμε να δούμε τι διατάξει μπορεί να είναι δεσμευτικές ή τι μπορεί να ισχύει κατά διακριτική ευχέρεια του υποκειμένου δικαίου παντού. Τώρα, για, να δούμε τώρα την επιστημονική διαδικασία Έχουμε σαφώς κάποια πρόοδο για φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό. Βλέπουμε εδώ πέρα ε, τι, τι διατάξεις ισχύουν άμεσα σε όλα τα κρατη και έτσι χαρακτηρίζουν την αγορά και το σύστημα το οποίο έτσι λειτουργεί. Ε, αυτά για το φυσικό Για τον ηλεκτρισμό τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα, αλλά τώρα έχουμε ε, ε, διάφορους, ε, διάφορα νομοθετήματα τα οποία ε, είναι έτοιμα προς, προς εφαρμογή. Άρα έχουμε θετικά μηνύματα από την εφαρμογή αυτή. Έχουμε τέσσερις χάρτες πόλης για τον ηλεκτρισμό, δύο φορτία χρονοδιαγράμματα και, κοιτάξτε, στο χάρτη αυτόν στη διαφάνεια. Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώνουμε ότι η αγορά λειτουργεί σε όλη αυτή την περιοχή που έχει το μπλε μοβ χρώμα από το, ε, από το μέχρι την ε, θάλασσα του Μπάρεντς. Οπότε και έτσι έχουμε βελτίωση των ροών της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό το είδους η σύνδεση των αγορών είναι πάρα πολύ βασική γιατί έτσι χρησιμοποιούμε τους διασυνδετές, τη διασύνδεση τέλος πάντων και είχαμε αύξηση αυτής της χρήσης της διασύνδεσης της διασυνοριακής 60% πήγε 77% σε τρία χρόνια για τον ηλεκτρισμό. Ακόμη έχουμε κάποιο πρόβλημα για κάποια είδους ροές. Τέλος πάντων, δεν είναι τα πράγματα τόσο ρόδινα όσον αφορά την αγορά intraday. Η, τώρα, η μακροπρόθεσμη μορφή, ε, της, η πτυχή της αγοράς, έχουμε εδώ πέρα περιφερειακή, περιφερειακής βάσης ρύθμιση, και όσον αφορά επίσης τον υπολογισμό της δυνατότητας παραγωγής έχουμε τη μέθοδο που βασίζεται στην ε, ροή. Όσον αφορά το φυσικό αέριο έχουμε εδώ πέρα διάφορα προγράμματα και έργα πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσον αφορά τη δυνατότητα διασύνδεσης. Βλέπετε εδώ πέρα τώρα το, το κόκκινο που είναι το πρίσμα αλλά έχουμε και άλλες περιφερειακές ε, αγορές και προγράμματα. Οπότε, βασικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα ε, προχωρούμε, αλλά υπάρχουν θέματα για τη σύγκληση των τιμών, κάποια προβλήματα, ε, επιπτώσεις των ανανεώσιμων στην αγορά. Πρόβλημα με το πώς θα υπάρχει σύγκληση και μείωση και πώς θα έχουμε κάποιο είδους ε, ε, περισσότερη ρευστότητα του, του κόμβου και πιο μακροπρόθεσμη ισχύ των διασυνδέσεων. Τώρα, όσον αφορά το ότι θα πρέπει να έχουμε ταχύτερη εφαρμογή του τρίτου πακέτου. Τους κώδικες οικοδικούς, τους ε, κόμβους που θα πρέπει να ε, τα καταφέρουμε σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τόσο διεξοδική παρουσίαση. Α. Ναι. Ε, είπατε ότι αυτή είναι η οπτική γωνία του οργανισμού, αλλά η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος του νομίσματος του οργανισμού είναι η όψη των ρυθμιστών. Και η δική σας ε, η θέση είναι και για μας άκρος σημαντική. Λόρδε Μόγκ, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Με, μου δίνει ιδιαίτερη τιμή το γεγονό ότι μου αποδίδεται τέτοια σημασία σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πραγματικά σημαντικό ότι ο οργανισμός χρησιμοποιεί εκπροσωπεί και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και τη συμβολή του στην όλη διαδικασία. Όπως βλέπετε, η Επιτροπή βλέπει ο οργανισμός να έχει επιτύχει καλά αποτελέσματα. Θα υπάρξει μια δεύτερη επίσημη αναθεώρηση την ερχόμενη χρονιά που ελπίζουμε ότι θα είναι εξίσου θετική. Πολύ σύντομα να αναφέρω εγώ ένα-δυο ζητήματα ακόμη που αφορούν περισσότερο τους εθνικούς ρυθμιστές. Σας αφήνω να διαβάσετε τα θέματα αυτά, αλλά ήθελα να σταθώ σε δύο συγκεκριμένα. Το δηλαδή την εμπορία ενέργειας και το bridge. Αυτά είναι τα τέσσερα θέματα του προγράμματος εργασίας μας ε, που έχουν ήδη προωθηθεί και που γύρουν βέβαια αρκετά ερωτηματικά. Το Γέφυρα για το 2025 λοιπόν. Τι ήταν αυτό το θέμα, το bridge. Αποφασίσαμε πριν από ένα χρόνο περίπου ότι ως ρυθμιστές θα λάβουμε μια στατικότερη τοποθέτηση για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον από ρυθμιστικής σκοπιάς στο ευρύτερο πλαίσιο που έχουν ορίσει τα θεσμικά όργανα. Θέσαμε το 2025 ως καταληκτική ημερομηνία γιατί είναι αρκετά μακριά αλλά όχι πολύ κοντά και λάβουμε υπόψη κάποια στατηγικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε την κοινωνία που δεν θα βασίζεται πλέον στον άνθρακα, τις μη προγραμματιζόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το αβέβαιο μέλλον για το αέριο, την ε, ε, ολοκλήρωση της αγοράς, αργό, βραδύτερη από ό,τι κάποιοι θα ήθελαν, όμως με νέους φορείς στην αγορά βλέπουμε ότι κατάλληλη έποψη εξασφαλίζεται και κάτι που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, το επίπεδο μελέτης, ε, το, η ομάδα μάλλον μελέτης ανώτερου επίπεδου ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνει κάποια έμφαση και στα θέματα της γειτονιάς μας, της ενεργικής γειτονιάς μας. Βλέπετε με γαλάζιο χρώμα τα συμπεράσματα που αντλήσαμε από τις προτάσεις. Να τονίσω ότι το τρίτο πακέτο είναι το απαραίτητο που πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να υλοποιηθεί από τα κράτη-μέλη και να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι κωδικοί. Θα πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με κατάλληλη διευθέτηση της αγοράς προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλουμε ιδίως προς την ε, ασφάλεια της παροχής αερίου και τη συνεργασία των εθνικών δικτύων. Βλέπουμε τώρα πόση σημασία έχει και ο καταναλωτής της ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο των πελατών, των καταναλωτών, δηλαδή να ενισχυθεί ο οργανισμός για να βεβαιωθεί ότι υπάρχει ρυθμιστική συνεργασία μεταξύ των ε, ενδιαφερομένων εδώ, ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τους υπευθύνους των δικτύων, ε, του συστήματος μετάδοσης, NTS και εδώ να υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία και συντονισμός. Τώρα το REMIT. Τι ήταν αυτό. Μετά από μια καταγγελία στις Ηνωμένε Πολιτείες είδαμε ξαφνικά ένα απλό ζήτημα καταγγελίας να παίρνει μεγάλες πολιτικές διαστάσεις. Εδώ βλέπουμε τι μπορεί να γίνει με ένα μικρό επεισόδιο για την εμπορία ενέργειας στην Ένωση γενικότερα τι διαστάσεις μπορεί να πάρει και αυτό ε, πραγματικά να απασχολεί ιδιαίτερος. Γι' αυτό τίθενται κάποια ερωτήματα βάσει του Ρήμικ. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά δεσμεύεται και ακολουθεί συνεπιστάσεις στο να πετυχεί μια ολοκληρωμένη διαφανή αγορά ενέργειας. Αυτό απαιτεί ότι θα εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών αλλά με την κατάλληλη ρυθμιστική στήριξη. Δεν ξέρω αν, Πρόεδρε, έχω χρόνο. Μήπως θέλετε εσείς, Διευθυντά μου, να συνεχίσετε με τις λεπτομέρειες. Διότι εδώ σας δίνω τις λεπτομέρειες του REMIT και το τι ακριβώς σημαίνει. Να σας δείξω μόνο τις διαφάνειες. Εντάξει, με μια ματιά. Βλέπετε ότι τα βασικά σημεία εδώ είναι Καταληκτική ημερομηνία Οκτώβριο 2015. Ε, λεπτομέρειες θα τις Με τις λεπτομέρειες θα καταλαβαίνατε καλύτερα, αλλά θα γίνουν σοβαρές αλλαγές τότε και του χρόνου θα υπάρξουν οι πρώτε καταχωρήσει. και σίγουρα τα πρώτα προβλήματα. Ο οργανισμό και οι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ ήδη ε, είναι προετοιμασμένε για τα προβλήματα. Τα δύο σημεία που είναι πολύ σημαντικά είναι το αυτόματο screening και η προκατακτική ανάλυση. Το πρόβλημα με την έλλειψη πόρων είναι κάτι που φαίνεται εδώ με τον πίνακα αυτό στο κόκκινο πλαίσιο, διότι χρειάζονται πολλοί πόροι για να γίνει σωστά η ανάλυση. Δεν μπορούμε να μετακινούμε ανθρώπους από τη μια υπηρεσία στην άλλη του οργανισμού. Χρειάζονται συγκεκριμένε δεξιότητες και προσόδα για το κάθε ε, ρόλο που αναλαμβάνεται. Αυτό είναι ένα μήνυμα, Πρόεδρο, που σας στέλνω εδώ Χρειαζόμαστε τους κατάλληλους πόρους, τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες, όχι μόνο στον Acer, αλλά και για τις εθνικές αρχές. Η συγκριτική αξιολόγηση και οι δείκτες της που ακολουθούνται παραμείως και στις ΗΠΑ και στο Βασίλειο δείχνουν ότι μεγάλους αριθμούς χρειάζονται. Και επίσης βλέπουμε τι πρόστιμα, τι κυρώσεις μπορεί να επιβληθούν ε, εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε πόσο μεγάλα ποσά. Βλέπετε εδώ το ποσοστό των ε, υποθέσεων που έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια και όπλες απλώ κοινοποιήθηκαν στον οργανισμό. Βλέπετε πω το επίπεδο ανεβαίνει και αυτή είναι απλώ η κορυφή του παγόβουνου. Ε, χωρί την κατάλληλη υλοποίηση, χωρί την απαραίτητη πρικοδότηση, υπάρχει πρόβλημα της, με τη φήμη, την αξιοπιστία του Acer για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ενεργειακή της Ένωση και για τα κρατη ενδεχομένω. Γι' αυτό πρέπει να δούμε πώς οι αρμόδιοι εθνικοί φωνείς, ε, φορείς θα στηρίξουν ε, αναλόγως την προσπάθειά μας, αλλά ε, βασιζόμαστε και στην αγαστή συνεργασία με την Επιτροπή σας, Πρόεδρε. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Ας περάσουμε στις δικές σας παρατηρήσεις κύριε Ευρωβουλευτές. Παρακαλώ. Ο κύριος Κόφορτ παρακαλώ. Πρώτος. Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας για, μια εξαιρετική, για τις εξαιρετικές σας παρουσιάσεις που υπογραμμίζουν κάποιες από τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν λέει ο κύριος Κόφορντ και η έκκληση για ιδίους πόρους που πολλοί από εμά η ανάγκη αυτή είναι κατανοητή λοιπόν από μας και σας ευχαριστώ επίσης για την έκθεση την παρακολούθηση της αγοράς. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και σημαντικά τα στοιχεία που απορρέουν από αυτό. Όπως γνωρίζετε, η εσωτερική αγορά ενέργειάς μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το μέλλον έχουν, έχει δύο νομίζω ξεχωριστά αλλά ξεχωριστές αλλά αλληλοσυνδεόμενες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η απόλυτη έλλειψη, έντονη έλλειψη επαρκών διασυνδετών και διασυνοριακά αλλά και μέσα στις ίδιες τις χώρες μας και τις ζώνες, τις ζώνες τους. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Θα ήθελα να τοποθετηθεί επ' αυτής. Δεύτερον, η διοργάνωση του αναγκαίου δυναμικού που ε, υφίσταται για παράδειγμα, πώς μπορεί να γίνει και η έκθεση παρακολούθησης της αγοράς νομίζω υπογραμμίζει αυτές τις προκλήσεις και στο τέλος τέλος κοστίζουν χρήματα όλα αυτά όταν δεν δημιουργούνται και δεν υφίστανται για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουν αυξηθεί οι τιμές ενέργειας ε, ηλεκτρικού σε όλες σχεδόν τις χώρες και αυτό αποτελεί πρόβλημα για τους Ευρωπαίους πολίτες σίγουρα. Αν μπορείτε να αποσαφηνίσετε περισσότερο πώς θα δράσετε για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και πιστεύω επίσης ε, Κάτι άλλο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε να αυξηθεί η συνειδητοποίηση, η ευαισθητοποίηση για αυτά τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε βέβαια, είναι θετικές οι εκθέσεις σας για αυτή την προώθηση, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, θα σας ήμουν ευγνώμων να το καταφέρναμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Πέτερσεν. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή που μας δώσατε. Αφενός τώρα, όπως γνωρίζετε καλύτερα από όλους, αυτά τα θέματα είναι πολύ ευαίσθητα. Τα κράτη-μέλη είναι πολύ ευαίσθητα στο να υπάρχουν υπερκρατικοί φορείς ε, που θα επιτηρούν και θα ε, προτείνουν και θα διοργανώνουν και το σχεδιασμό και τα συναφή η ειλικρινή άμεση ερώτηση προς εμάς που γνωρίζω ότι θα θεωρήσετε αδύνατο να απαντήσετε ειλικρινά. Η ερώτηση είναι βρισκόμαστε εκεί όπου θα θέλαμε να βρισκόμαστε όσον αφορά τη διακυβέρνηση και διαχείριση. Διότι στην καθημερινή σας δουλειά θα πρέπει να αντιμετωπίζετε πολύ μεγάλες δυσκολίες όταν έχετε απέναντί σας εθνικούς φορείς ε, προωθώντας ε, την διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία διασυνοριακά. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Αν θέλουμε να πετύχουμε την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση και αν χρειαζόμαστε, αν θέλουμε να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται μεγαλύτερη, περισσότερη συνεργασία σε όλα αυτά και συντονισμό. Σύντομη ερώτηση λοιπόν προ εμά. Βρισκόμαστε εκεί όπου θα θέλαμε να είμαστε όσον αφορά τη διακυβέρνηση και διαχείριση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο Τούρμε, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Καθυστέρησα, αλλά όντα στην αίθουσα κάπου, κατά κάποιο διάστημα γνωρίζω περίπου περί τίνο πρόκειται. Για το Remit Λοιπόν, από κοινού ρυθμίσαμε, κάναμε τα προαπαιτούμενα για αυτό το νομοθετικό έργο και πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη. Αν απολεστεί η εμπιστοσύνη χαθήκαμε, θα βρεθούμε σε μια δραματική κατάσταση πραγμάτων. Και θα έλεγα ότι ακριβώς ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις. Έχετε λάβει κάποια θέμα περιπτώσεις σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Πείτε μας δύο λόγια για το ποια είναι η διαδικασία ανάλυσης όλων αυτών και πώς συνδέονται σε σχέση με τα θέματα των οποίων επιλαμβάνεστε. Διότι γνωρίζουμε ότι θα θέλατε να υπήρχαν περισσότερα στελέχη. Αν θα μας λέγατε όμως γιατί ακριβώς χρειάζονται περισσότερα στελέχη να σας βοηθήσουν, αυτό ίσως θα ήταν κάτι το επικοδομητικό. Ένα άλλο που θα ήθελα να υπογραμμίσω ως θέμα είναι η διαφορά μεταξύ των χονδρικών τιμών αγοράς και λιανικών τιμών αγοράς. Η διαφορά αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό στο ETS, στο ETS. και αν υπάρξει μια, ε, τέτοια, ένα τέτοιο πρόβλημα πώς μπορούμε να αναμείνουμε να ανακάμψει και να βελτιωθεί η κατάσταση σε σχέση με την αγορά. Οι τιμές ε, θα πρέπει να δούμε ότι θα παραμείνουν ως έχουν. Αυτό το οποίο προτείνεται και λέτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είσαστε εκφράζετε τη θλίψη σας για αυτά τα χαμηλά ποσοστά. Θυμάμαι όμως ότι το 2003 όταν ήμουν εισηγητής για αυτήν την οδηγία η δική μου πρόβλεψη ήταν ότι οι καταναλωτές δεν θα πάνουν ώρες, ατέλειωτες ώρες για να εξεύρουν αν θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν κάποια λίγα χρήματα. Νομίζω είναι αυταπάτη. Ένα, μια σήμερα, ένα χειμερικό όνειρο ότι οι πολίτες, οι καταναλωτές τελικά ότι το switching, η διασύνδεση ξαφνικά θα αυξηθεί δραματικά όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ αυστηρότερη νομοθεσία. Και αυτό που κάναμε στην αγορά τηλεπικοινωνιών, γνωρίζαμε ότι υπήρχε εξαπάτηση των πολιτών στη λιανική αγορά εις βάρος των καταναλωτών. Τι κάναμε σε σχέση με τις τιμές ρυθμίσαμε πλαίσια και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε σκληρά, αυστηρά μέτρα διότι πώς μπορεί να εξηγήσει κανείς σε σχέση με τις τιμές αγορών πώς μετατρέπονται και μεταφράζονται σε χαμηλές τιμές, χαμηλότερες τιμές στη λιανική αγορά και που δεν μπορούν να αγοράσουν με υποφελή τρόπο από τους ε, ε, εμπόρους ε, σε ευνοϊκές τιμές. Χρειάζονται λοιπόν αυστηρότερες. Ο κύριος Ηλικιώτης παρακαλώ έχει τον λόγο. πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίαση που είχαμε από τον κύριο Ποδόσιν και τον Λόρτ Μοκ. έχει επιτελέσει ένα σημαντικό έργο στα τρία χρόνια λειτουργία του ΑΣΕΡ Ωστόσο, ε, προβάλλεται συνεχώς ένα στόχος για περιττέρω ενίσχυση των εξουσιών σε κεντρικό ε, ε, επίπεδο, δηλαδή μεταφορά εξουσιών από εθνικές ανεξάρτητες αρχές στη διεδοκισία του Άσερ. Και στο βαθμό που είναι ισοπεδωτική και αδεικμηρεί ότι όχι μόνο θα ωφελέσει αλλά μπορεί να καταστρατηγήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών σε αντίθεση με τι είπε ο προηγούμενος ο ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν τα κράτη, ο κρατικό έλεγχο στη ρύθμιση ενεργειακή αγορά σε εθνικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν πρέπει να παραγνωρίζεται. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω όμω του ε, ε, αξιότιμου ομιλητέ μα, εκπροσώπου του ΑΣΕΡ, ποια πλειονεκτήματα ή μειονεκτήματα βλέπετε να προκύπτουν από τη μεταφορά του ελέγχου της ενεργειακής αγοράς σε κοινοτικό πλαίσιο πάνω από τα εθνικά ρυθμιστικά προγράμματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, Σας ευχαριστούμε, Βαν Νιβενχόιζεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ρωτήσω κάτι όσον αφορά από πλευράς τη ρυθμιστική πλευρά του νομίσματος όπως είπατε και εσείς για το Ρέμετ γιατί στις, ε, στις αναφέραμε τις έρευνες για κατάχρηση της αγοράς, για χειραγωγήσεις κλπ. Και θα ήθελα επίσης να ρωτήσω σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν για παγκόσμια κριτήρια, ορόσημα, δείκτες κλπ. Τα benchmarks. Εσείς πώς θεωρείτε ότι αυτός συντεριάζει και συμβαδίζει και συνάδει με το Ρίμιτ. Πώς συνδυάζονται αυτά όλα. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα από αυτού. Ευχαριστώ. Μπούζεκ, σας ευχαριστώ κυρία. Κυρία Καμπεθόν Ρουίς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα ευχαριστούμε τους ε, συγκητές και τους δύο. Συγκεκριμένο ερώτημα τη γνώμη τους για κάτι που έγινε στη χώρα μου. Πρόσφατα, όπως ξέρετε, στην Ισπανία, στα πλαίσια κάποιων μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων, είχαμε συγκέντρωση και συγχώνευση ρυθμιστικών αγορών για τηλεπικοινωνία, ενέργεια κλπ. και επίσης των ταχυδρομείων. Και έχουμε τώρα τη συγκεκριμένη επιτροπή για, την, ε, για, για τον ανταγωνισμό. Είχαμε επομένως κάποιες αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση και έχουμε επομένως τώρα το καινούριο καταστατικό, το καινούριο νόμο που θα διέπει αυτές τις ε, υπηρεσίες, αυτούς τους τομείς. Εσείς αυτές τις αλλαγές που έκανε η κυβέρνηση πώς τις αξιολογείτε. Ράμστορφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω τρεις ερωτήσεις. πρώτο πρώτο Στο παρελθόν, τότε που ετοιμαζόταν η τρίτη δεσμέτρων για την ενέργεια, ε, είχαμε ο πλευράς Μόργαν την έννοια της ενεργειακής φτώχειας. Τι γίνεται με το πρόβλημα της ισότητας πρόσβασης στην ενέργεια πανευρωπαϊκά. Διότι σε κάποια κράτη, σε κάποιες περιοχές αυτών είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση στην ενέργεια. Έτερον, γνωρίζουμε εμείς που εργαζόμαστε ε, αρκετό και σε αυτή την Επιτροπή, όπως και ο αξιότιμος πρόεδρός μας, ότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις όσον αφορά τον συντονισμό των εθνικών Εθνικών αρχών, όπως κάποια παρέκκληση για την Γερμανία. Εξαίρεση για τον συντονισμό των εθνικών αρχών και είχαμε αποκρισταλώσει συγκεκριμένη θέση. Μου είπαν ότι αυτό δεν ισχύει, δεν ξέρω εσείς μπορείτε να μας ε, ξεκαθαρίσετε για το ότι κατηργήθησαν αυτές οι παρεκκλήσεις και εξαιρέσεις. Τρίτη παρατήρησή μου, Ενεργειακή Ένωση. Αναφέρθηκε και είναι κάποια ιδέα που κυκλοφορούσε στο παρελθόν, ε, κύριε Μπούζεκ εσείς. Έχουμε τώρα επίτροπο αρμόδιοι για την Ενεργειακή Ένωση και φαντάζομαι κάτι έχετε να μας πείτε όσον αφορά αυτήν την ένωση. πέστε μας την άποψή σας. Uh, Μπούζεκ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητεί άλλο το λόγο. Όχι, από ό,τι φαίνεται επομένω. Και τώρα να αρχίσουμε τις απαντήσεις από τους εκπροσώπους των ρυθμιστικών αρχών. Έχει το λόγο κύριε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ τεκμηριωμένες οι ερωτήσεις, οι παρεμβάσεις. Με τα γενικότερα θέματα πρώτα. Με το ερώτημα του κυρίου Πέτασε να ξεκινήσω για τη διακυβέρνηση διαχείριση. Αυτό ήταν το κεφάλαιο που περισσότερο απασχόλησε τους εκπροσώπους των πολλών εμπλεκομένων σχετικά. Ξεκινήσαμε με αυτό που νομίζουμε ότι είναι επιτυχία αν κάτι δεν έχει σπάσει τότε μην προσπαθήσετε να το επισκευάστε. Και νομίζω ότι οι ρυθμιστές για τον οργανισμό και για τις εσωτερικές δομές όσον αφορά τους ελέγχους και τις ισορροπίες ήταν πολύ αποτελεσματική η προσπάθεια ως εγχείρημα. Η πρότασή μας είναι να μην προσπαθήσουμε να άρουμε ή αλλάξουμε κάτι σε σχέση με το μηχανισμό αυτόν όπως λειτουργεί σε σχέση με τα διάφορα στοιχεία, το επιδιαιτητικό ε, σκέλος, ε, το ε, εκτελεστικό και τους κανόνες για τη διαφάνεια. Ωστόσο πιστεύουμε επίσης εξίσου ότι μεγαλύτερη διακυβέρνηση και μεγαλύτερο πλαίσιο διαχείρισης χρειάζεται για συγκεκριμένα θέματα. Εκείνα τα οποία συνενώνουν τις ρυθμιστικές αρχές. Όχι επειδή θεωρούμε ότι κάτι το αρνητικό ή κακό υπήρξε, αλλά επειδή αναγνωρίζουμε ότι είναι πιθανότατο ότι ο όγκος εργασίας που θα έχουν αυτοί οι φορείς στο μέλλον θα αυξηθεί. Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε ο οργανισμός, η υπηρεσία θα έχουν τους πόρους να τα αντιμετωπίσουν όλα μόνοι τους. Γι' αυτό υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη, όπως το βλέπουμε εμείς, για να υπάρξει η σωστή ρύθμιση και λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρούμε ότι πρέπει να ε, εξεταστεί αυτό. Είναι ανάγκη να το εξετάσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να τα αποκριθούμε. Τρίτον, έχει τον τίτλο η ε, οργάνωσή μας ε, την λειτουργία, την λειτουργικότητα. Και γι' αυτό αναγνωρίζω μεγαλύτερο πλαίσιο άτυπης συνεργασίας που θα λειτουργεί όχι μόνο μέσω του οργανισμού αλλά και μέσω των άλλων οργάνων μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών επίσης. Πριν από δύο χρόνια όταν προσήλθα για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιμετώπισα την κατάσταση εκεί, είχαμε πολύ λίγες επαφές με τους άλλους συναδέλφους. Δεν ήταν καθαρά βρετανικό πρόβλημα αυτό. Οι περισσότεροι, εκτός αν ήταν σε περιφέρειες, είχαν πολύ λίγες επαφές μεταξύ τους. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Υπάρχουν επαφές που έχουν θεσπιστεί με περιφερειακούς φορείς και τομείς και η υπηρεσία γενικά είχε καλές επιδόσεις. Μπορεί να βελτιωθεί, αλλά οι επιδόσεις ήταν γενικά θετικές ήταν αποτελεσματική. Θα έπρεπε να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τα θέματα διαχείρισης και διακυβέρνησης και πάλι πιστεύω ότι η διαφάνεια των στοιχείων πληροφόρησης και για την αγορά και για το πλαίσιο δεκαετούς ανάπτυξης και για τις προοπτικές του αφορά το χειμώνα για παράδειγμα μας δίνει μια πολύ καλύτερη εικόνα για την Ευρώπη. Τα πράγματα και πάλι εδώ βλέπουμε βελτιώνονται. Και ένα τελικό παράδειγμα στις υποδομές, στην ανάπτυξη του πακέτου υποδόμων της δέσμης μέτρων για τις υποδομές όπως αναφέρατε. Καταφέραμε να αναπτύξουμε σε στενή συνεργασία <clears throat> με μικρό πλαίσιο υποστήριξης νομοθετικά αλλά με μεγάλο πλαίσιο ανάλυσης ε, και εμβάθυνση στο τι θα μπορούσε να γίνει ως προοπτική στο μέλλον. Αυτό που θα γίνει στο μέλλον, η προσωπική, προσωπική άποψή μου είναι ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ολοκλήρωση από πλευράς της υπηρεσίας μας. Υπάρχει ήδη μεταξύ των συμβαλωμένων μερών ένα πλαίσιο μηχανισμού επίλυσης ε, ε, επιμάχων θεμάτων. Θα υπάρξει λοιπόν μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Μια ολοκληρωμένη αγορά θα το απαιτήσει αυτό. Η αποτελεσματικότητα θα απαιτήσει μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης. Και αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή είναι η απάντησή μου στην πρώτη παρέμβαση. Στην δεύτερη, τρεις τώρα παρατηρήσεις. Ε, παινία ενεργειακή. Πρέπει να δούμε την ουσιώδη διαφορά μεταξύ του βορρά της Ευρώπης των σκανδιναβικών χωρών όσον αφορά την ενεργειακή παινία ξεχωριστά για αυτές τις χώρες αντί για ένα γενικά κοινωνικό πρόβλημα για όλους. Και πάλι προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει ένας πολύ καλύτερος τρόπος. Η ενεργειακή παινία δεν είναι ένα πρόβλημα ποσοστού που δαπανάτε για, την, ε, ε, για τα ενεργειακά. Είναι το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από συγκεκριμένες χώρες. Έχουμε αυτό το θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από πλευρά μας που θέτει διαφορετικές προκλήσεις μεταξύ ενός ενός ε, του χειμώνα στο βορρά και ενός υπιότερου χειμώνα στην Πορτογαλία, στην Ισπανία ή στις άλλες χώρες του Νότου. Συνειδητοποιώντας αυτά και αυτό πάλι αφορά τη δική σας παρέμβαση θα μπορέσουμε να δούμε κάποια βελτίωση σχετικά. Όσον αφορά τώρα για, τους, ε, για την εξαίρεση που ρωτήσατε, το Βίλνιους είναι πλήρως εμπλεκόμενο ε, στοιχείο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο διασφαλίζεται η ανεξαρτησία λειτουργίας. Τρίτη ερώτηση. Είναι πρόκληση για μένα να απαντήσω. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα το τι θα μπορούσα να απαντήσω. Η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει κάποια από τα θέματα τα οποία τίθενται. Ένα από αυτά τα θέματα είναι και αφορά και την παρατήρηση του Προέδρου για την ενεργειακή κοινότητα που πρέπει να δημιουργηθεί. Αυτό θα έχει κέρια σημασία εμείς με τους περιορισμένους πόρους μας προσπαθήσαμε να σημειώσουμε πρόοδο, να προχωρήσουμε και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις δραστηριότητες της Ένωσης με την κατάρτιση και εκπαίδευση ε, υπαλλήλων. Αυτό θα είναι ένα δραστήριο μέρος, μέρος των εργασιών μας. Μια ολοκληρωμένη αγορά θα βρίσκεται στον πυρήνα αυτών των δραστηριοτήτων και θα ενδυναμώσει, θα ενισχύσει τις προσπάθειες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ακούσαμε και από προηγούμενες παρεμβάσεις. Σε σχέση με τη δική σας παρέμβαση όσον αφορά την ισπανική κατάσταση, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια δεδομένη, κομμένη και ραμμένη απάντηση. Οι νέες ε, διατάξεις, ε, οι νέοι κανονισμοί όπως στην Ολλανδία και σε άλλες χώρες που εξετάζουν αυτές τις μικτές ε, ρυθμίσεις η νομοθετική αυτή προσπάθεια συνεισφέρει θετικά στο έργο μας και είναι πολύ ενδιαφέρουσα συνιστόσα και έχουν και βιώματα από το πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών. Οι δύσκολες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν από τον Διευθυντή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Τώρα έχετε εσείς τον λόγο να τοποθετηθείτε, κύριε Ποτότσνικ. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις και επίκαιρες. Επιτρέψτε μου να τις πάρω σε σχέση με το REMIT πρώτα, να δούμε εκεί δηλαδή που βλέπουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση. Εσείς ε, κύριε Κόφαρ, μιλάμε για α, κομβικούς ε, συνδετήρες, σημεία σύνδεσης πόσο ικανοί είμαστε το δυναμικό αυτό να διασφαλίσουμε ότι θα υφίσταται και θα χρησιμοποιείται με τον καλύτερο βέλτιστο τρόπο. Σίγουρα πιστεύω ότι θα έχετε συνειδητοποιήσει και θα γνωρίζετε ότι όταν έχουμε το θέμα ανάπτυξης δυναμικού για τη διασύνδεση υπάρχει ένας νέος κανονισμός όσον αφορά την ε, ε, μετάδοση, την μεταφορά ενέργειας στην Ευρώπη και είχαμε τον πρώτο γύρο για τα προγράμματα κοινού συμφέροντος που είναι η απάντηση θα λέγα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πρόβλημα που πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει υποδομή αναγκαία εκεί όπου χρειαζόμαστε με προγράμματα προτεραιότητας που θα υποφεληθούν από μια ολόκληρη σειρά από προτερήματα που θα δημιουργούνται. Και αυτό είναι για μια συγκεκριμένη περίοδο η κατανομή του κόστους και πιθανότατα και η πρόσβαση και όλα στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που θα διασφαλίζεται. Αλλά πιο βραχυπρόθεσμα, αμεσότερα, διότι αυτό απαιτεί χρόνο το άλλο που περιέγραψα, θα πρέπει να μας κάνει να δράσουμε με τον βέλτιστο τρόπο και στην η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρισμού, καταφέρνουμε με την, τα έργα μας, με τις προτεραιότητές μας να, να ανταποκριθούμε και ίσως θα μπορούσαμε να δούμε στην οθόνη την αντίστοιχη σελίδα. Εδώ βλέπουμε πώς ε, το market capping που δεν λειτουργεί ακόμα, πώς η ροή του, ε, του προϊόντος της, ε, του ηλεκτρισμού ακολουθεί συγκεκριμένη πορεία. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι 30% αυτό. 50% διορθώνει 30 ή 40%. Αλλά αν δείτε στο άκρο δεξιά της διαφάνειας του γραφήματος έχουμε το όριο μεταξύ Ουγγαρίας και Σλοβακίας και έχουμε μηδενικό επίπεδο στο 2013. Γιατί κατάφερε η ενέργεια να ρέει με τον σωστό τρόπο. Επειδή εισήχθη το market capping σχετικά το 2012 και αυτό είχε αυτό το αποτέλεσμα. Μπορούμε δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να είμαστε ε, αποτελεσματικοί. Και αν δούμε το επόμενο γράφημα, την επόμενη διαφάνεια, θα δείτε ποια, ε, τι ισχύει για την κοινωνική ευημερία και ποιες επιπτώσεις υπάρχουν σήμερα επειδή δεν χρησιμοποιούνται με τον σωστό τρόπο interconnectors, οι, διασύνδε, οι διασυνδέσεις. Μπορώ να δώσω και άλλα παραδείγματα. Είναι σαφώς προτεραιότητα για μας στο, στον επιμερισμό δυναμικού για το φυσικό αέριο. Ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Γι' αυτό θέλαμε να έχουμε εθελοντικό πλαίσιο εφαρμογής. Διότι αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε έτσι πολύ ταχύτερα να αντιμετωπιστεί από ότι αν ακολουθούσαμε κανόνες, διατάξεις κανονισμούς που επίσημα θα έπρεπε πρώτα να εγκριθούν και μετά να υλοποιηθούν. Χονδρικές και λιανικές τιμές του κυρίου Τούρμες. Ναι, πράγματι και εμάς μας προβλημάτισε αυτό. Ήταν ένα ένιγμα, ένα πρόβλημα. Έχουμε δυσδιάστατη κατάσταση εδώ. Υπάρχει διασύνδεση μεταξύ κάποιου προϊόντος στις τιμές χονδρικής στις τιμές λιανικής και στο συσχετισμό τους με τις τιμές χονδρικής πώς συνδέονται και συσχετίζονται. Είδαμε ότι δεν ισχύει παντού αυτός ο συσχετισμός, αυτή η αναλογία. Και αν μπορούμε άμεσα να περάσουμε σε μια διαφάνεια που έχω εγώ εδώ, θα δείτε ότι σε κάποιες χώρες αυτός ο συσχετισμός λειτουργεί ομαλά και καλά και κάτω μπορείτε να δείτε ότι η συνιστόσα για αυτές τις ενεργειακές ε, τιμές ε, μεταξύ ε, χονδρικής και λιανικής συσχετίζονται, αλλού όμως όχι. Σε άλλες χώρες όχι. Αυτή είναι η πρώτη πτυχή που θα έπρεπε να δημιουργήσει κάποια ανησυχία, κάποια μελήματα. Και αφορά ίσως θέματα ανταγωνισμού αυτά. Μετά όσον αφορά το συνολικό, τη συνολική τιμή ηλιανικής, και είπα ότι ε, το, η συνιστόσα της ενέργειας είναι ένα μικρότερο ποσοστό, λιγότερο από 50% της τελικής τιμής, θα, ανέβαινε, θα ανέμενε κανείς ότι αυτός ο συσχετισμός θα ε, απεσβαίνεται, θα χανόταν στο τέλος γιατί έχουμε μια πολύ μικρή ε, συνιστόσα στις ε, τιμές που αντανακλούν το κόστος ενέργειας. Τώρα, για το switching. Και αυτό μας ανησυχεί, μας δημιουργεί κάποια προβλήματα όταν υπάρχουν κιόλας και σημαντικές εξοικονομήσεις που μπορούν να επιτευχθούν. Αναφέρομαι στη διαφάνεια 47 τώρα. Εδώ προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ των εξοικονομήσεων που μπορεί να επιτευχθούν με το switching και το ποσοστό switching μπορούμε να δούμε θετικές επιπτώσεις όσον αφορά την επίπτωση στο φυσικό αέριο. Εδώ βλέπουμε σε σχέση με τις εκτιμήσεις μας εκατοντάδες ευρώ μπορούν να εξοικονομηθούν με το switching, με την μετατροπή αυτή. Και όμως δεν μετατρέπουν οι καταναλωτές. Θα προσπαθήσουμε να μεγεθύνουμε την εξέταση αυτού του προβλήματος σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες και θα γνωρίζουμε περισσότερα το 2015. Για τον κύριο Σιλικιώτη, εσείς κύριε εκφράσατε ανησυχία και σας προβλημάτιζε ο ρόλος της ευρωπαϊκής διάστασης ε, όσον αφορά θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα. Πρέπει να σας πω ότι η πορεία νομίζω δεν είναι καμιά άλλη παρά μεγαλύτερη, μεγαλύτερο εξευρωπαϊσμό όλων των ε, παραμέτρων του ενεργειακού τομέα. Αυτό μπορεί να δώσει πολύ μεγαλύτερη ε, προώθηση και όσον αφορά και τον, ε, την αρχή, την, τον οργανισμό μας, αλλά ακόμα και με εμπλοκή των εθνικών ε, αρχών. Και εδώ πρέπει να βρούμε μια ευρύτερη συνταγή για ευρύτερο συντονισμό και συνεργασία στο ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ όλων. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στη συνέχεια στο remit και πάλι, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το άφησα για το τέλος, στην τελική μου παρέμβαση. Για περιπτώσεις ρωτήσατε. Ναι, ήδη παίρνουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις και επιλαμβανόμεθα αυτών. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το νέο πλαίσιο εποπτείας παρακολούθησης που να λειτουργεί ήδη, να είναι λειτουργικό. Είναι έτοιμο. Το σύστημα αναπτύχθηκε, εκπονήθηκε κατά τα τελευταία δυόμιση έτη. Ωστόσο, η υποχρέωση καταχώρησης ε, αυτών των περιπτώσεων και στοιχείων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2015 το αργότερο. Όμως ε, σε σχέση με το ε, REMIT και την έναρξη κατά το 2011 το Δεκέμβριο περιπτώσεις που αναφέρονται από συγκεκριμένα θέματα αγορών, συγκεκριμένους εμπλεκόμενους αγορών αλλά επιλέγονται, συλλέγονται από εμάς σε ένα επίπεδο ad hoc ε, εκ των ενόντων, αλλά σε άλλες περιπτώσεις έχουν αυξηθεί περιπτώσεις ε, κατά, κατά τη διάρκεια του 2014. Πάνω από 50 περιπτώσεις έχουν γνωστοποιηθεί σχετικά σε εμά. Υπάρχει ίσο ποσοστό όσον αφορά την πληροφόρηση, την εκ των ένδων πληροφόρηση σε επιχειρήσεις και ε, ρόλο ε, καταχρηστικό στις αγορές καταλήξαμε στο ότι υπήρχε παραβίαση ενός από τους όρους του Ουρίμιτ. Πώς αυτό τώρα έχει επιπτώσεις ε, στους, ε, στους πόρους μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε 30 περιπτώσεις ετήσια χοντρά χοντρά. Έχω εδώ 6 στελέχη, 6 άτομα αυτή τη στιγμή. Αν ε, θέλαμε να το κάνουμε αυτό διαζώσει ζωντανά, μόνο έξι στελέχη θα μπορούσα να επιμερίσω. Αυτή τη στιγμή όμως 2 στελέχη έχω μόνο διότι οι άλλοι προσπαθούν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες ε, ε, ολοκλήρωσης λειτουργικών διατάξεων για τη λειτουργία του REMIT. Η δική μου εκτίμηση ποια είναι. Θα χρειαζόμαστε κάπου 20 με 25 περισσότερα άτομα στελέχη για να κάνουμε αυτή τη δουλειά σωστά και έχει υποστηριχθεί αυτή η εκτίμησή μου από το σώμα των ρυθμιστών, το, σώμα των ε, ε, εκπροσώπων των ρυθμιστικών αρχών. Και αυτό σε σχέση με μια ανάλυση έργου, αν θέλει κανείς ε, να το δει, υπάρχουν σελίδες επί σελίδων περιγραφής συγκεκριμένου έργου για να μπορέσει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά το REMIT μέσα στο πλαίσιο και των απαιτούμενων πόρων που θα χρειαζόμαστε. Όλα αυτά ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με αυτά που άλλοι φορείς ε, και ε, υπεύθυνοι για τέτοια θέματα χρησιμοποιούν ή εκτιμούν αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η πρόκληση λοιπόν. Δεν θα είμαστε σε θέση, δεν θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις κατεπηγόντων ε, που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με τα θέματα εμπορίου και συγκεκριμένων στοιχείων. Αυτή τη στιγμή πάνω από μισό εκατομμύρια τέτοια στοιχεία θα υπάρχουν. Εκτιμούμε ότι θα υπάρξουν πάνω από ένα εκατομμύριο. Δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους όγκο μεγεθών με, με λίγα στελέχη ακόμα και σε ένα καλό ε, σύστημα. Ε, θα πρέπει να εντοπίζουμε τις ε, ανομαλίες, ε, τα έκτακτα περιστατικά και εκεί ακριβώς μπορούμε να πούμε ότι αυτό θα είναι το ουσιοδέστερο. Τώρα, αυτό αφορά μεταρρύθμιση, αναθεώρηση των benchmarks, των βέλτιστων προδιαγραφών. Είναι προφανές ότι υπήρξε κατάχρηση της εφαρμογής των βέλτιστων προδιαγραφών, αλλά υπάρχει και κάτι παραπάνω από αυτό πίσω από αυτή την ιστορία. Θα βοηθούσε να είχαμε νέους κανόνες και κανονισμούς, αλλά αυτό είναι μόνο μικρό μέρος του προβλήματος που ρυθμίζεται έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ, ε, Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε πάλι το λόγο, αλλά δεν θα ήθελα να σας μιλάω για λεπτομέρειες και όχι για το γενικότερο, το σημαντικό θέμα. Η εκτίμησή μας από το Συμβούλιο των Ρυθμιστών και από τον ίδιο το Διευθυντή είναι εκτιμήσεις πολύ ψηλότερε από αυτές που υποβάλλει για την ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για την ώρα βρισκόμαστε σε φάση προγράμματο εργασία που δεν θα ολοκληρωθεί πριν εγκριθεί και ο προπολογισμό στο τέλο τη χρονιά. Αλλά αυτό που εννοούμε και λέμε προ την Επιτροπή σα, καθώ δεν είναι εκείνη που θα αποφασίσει για τον προπολογισμό, αλλά στο παρελθόν έχει στηρίξει, δείχνοντα κατανόηση για τι δυσκολίε ε, του οργανισμού μα, είναι άποψη όλων μας ότι μπορούμε να μετατοπίσουμε πόρους και να διαχειριστούμε τη διαδικασία όπως προβλέπετε από το REMIT. Ιδάλλως θα έχουμε σοβαρούς τριγμούς του χρόνου. Συνάδελφοι, πραγματικά ε, οι βουλευτές πρέπει να το έχουν αυτό υπόψη τους και οι ρυθμιστικές αρχές όταν λαμβάνουν την απόφαση αυτή όταν λάβουν την απόφαση αυτή του χρόνου. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να πάει και στους συναδέλφους εδώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους προσκεκλημένους μας για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσαν. Ε, ε μας δώσατε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την Επιτροπή μας. Μία είδηση για σας. Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας επαφής Άσερ με εκπροσώπους από την Άσερ, τους δύο προσκεκλημένους μας δεύτερη εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Στις 9 Δεκεμβρίου μάλλον. Προς επιβεβαίωση. Αλλά 9 Δεκεμβρίου. Πολύ σημαντική ημερομηνία για τα μέλη της ομάδας επαφής Άσερ από την Επιτροπή Ήτρε. Πρέπει να διατηρήσουμε στενές επαφές και αν μου επιτρέπετε θα σας ευχαριστήσω για την επίσκεψή σας στην Επιτροπή Ήτρα. Δεν είναι καθόλου η τελευταία φορά. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως το τι γίνεται με την ομάδα επαφής και τους 16 συναδέλφους, όσους συμμετέχουμε εκεί, αλλά και όλους τους υπόλοιπους, τα μέλη της Επιτροπής μας. Εσωτερική ενεργειακή αγορά, θέμα άκρα σημασίας για όλους μας, για την ευρωπαϊκή ενεργειακή κοινότητα. Πριν από λίγου μήνες ξεκινήσαμε να λέμε για ενεργειακή κοινότητα, τώρα λέμε για ενεργειακή ένωση. Πάρα πολύ σημαντική ιδέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα δημιουργήσουμε ένα νέο φορέα από το πουθενά με δικού της διοικητικού πόρου. Αλλά είναι μια ιδέα πολύ ε, έξυπνη, πολύ ε, εύστοχη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Συνάδελφοι, πολύ καλά νέα για σας. Αύριο στις 9 το πρωί, τρίτο μέρος της συνεδρίασής μας και τώρα η συνεδρία των συντονιστών. Οπότε άλλη μια ώρα για τους συντονιστές μας. Σας δίνω τρία με πέντε λεπτά διάλειμμα για να μείνουμε και μόνοι σε αυτή την αίθουσα. Συγγνώμη που το θέτω έτσι.